Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Δεν θέλω να καθυστερούμε άλλο. Ε, πολλοί ε, άφησαν την κάρτα τους και εγώ, συμπεριλαμβανομένου. Ε, αφήσαμε την κάρτα της ψηφοφορίας στην άλλη αίθουσα. Ε, οπότε, εντάξει, θα χρειαστεί λιγάκι ο γραμματέας να, μετρά, να μετράει χέρια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. So, uh, Mr. Engstrom, our Η συγκέντρια είναι εδώ. Συγγνώμη που δεν μπορούσαμε να, το, να δούμε την έκθεση σας ε, σήμερα. Μήπως, ε, το πρωί δηλαδή, μήπως θέλετε να πείτε κάτι πριν να ψηφίσουμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τους σκιώδες και τη γραμματεία. Δύο συναντήσεις κάναμε. Πολύ χρήσιμες, πολύ επικοδομητικές. Οπότε ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Δεν έχω να πω εγώ τίποτα άλλο. Okay, Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Οπότε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Uh, uh, τροπολογία 2 που θα προσθεθεί ως νέα προ... παράγραφος. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αποσύρεται η τροπολογία της κυρίας Κόμη. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε μια συμβαστική τροπολογία. Γκέπχαρτ και κόμι. Ψηφίζουμε. Υπέρ τη συμβαστική πρόταση. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 6 και 13 καταπίπτουν. Πάμε στην 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Ζιβάν και, καβαλα... και καβαντά. Υπέρ. Κα... Υπέρ. Μάλλον να μετρήσουμε πρέπει. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. You It's 11 11, 12. okay, defeated by one vote. Ε, απορρίπτεται για μία ψήφο. Τα μέλη της Επιτροπής που δεν έχουν ε, ενημερώσει την γραμματεία και ψηφίζουν, πείτε το, ε, πρέπει και τα μέλη των υπολείπων επιτροπών πρέπει να στείλουν ένα ε, σημείωμα στην γραμματεία που τους ορίζει η ομάδα τους αν θέλουν να ψηφίσουν. Σας το θυμίζω. Τροπολογία 9. Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δέκα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έντεκα, Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Δώδεκα.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 να θυμίσω ότι μόνο τα μέλη της Επιτροπής μας μπορούν να ψηφίσουν, εκτός αν έχουν ενημερώσει την γραμματεία. Ποιος είναι υπέρ για τη συμβαστική τροπολογία 2. Και ξαναμετράμε βέβαια. Okay. Um, Ποιος είναι κατά? Okay, is 18 to 10, okay. Εγκρίνεται. 18 προς 10. 14 και 15 καταπίπτουν. Πάμε στην τροπολογία της κυρίας Κόμη, 16 με προφορική τροπολογία που τη βλέπετε στο έγγραφο. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16 καταπίπτει. 18 του Ζουβάν υπέρ. Για μια διαγραφή πρόκειται εδώ. Ποιος είναι υπέρ. That's 19 in favor against... 19 υπέρ. Ποιος είναι κατά. Okay. Okay, that's 10 against. Amendment 17 uh, falls. Η 17 καταπίπτει. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Those against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 και 20 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα για την έκθεση. Ποιο είναι υπέρ. Και κρατήστε τα χέρια σα ψηλά για να μπορέσουμε να μετρήσουμε. Κατά. Είναι κανεί κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ποιο είναι κατά. Α, να, είναι και ένα κατά. Πρέπει να μετρήσει τώρα πώ είναι υπέρ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια στον Κρίστιαν Έγκστρομ για την πρώτη σας συγχρηματοδότηση. Αναμένουμε λοιπόν και τις επόμενες. first time in this room. Yeah. It's a new. The other you come you did your hearing in here. It's a hearing in this room. Yeah. First time. so um, I can just say good afternoon, everybody, to those. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην τελευταία συνεδρίασή μας για αυτό το μήνα. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να καλωσορίζω τον Επίτροπο Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, τον Αντώνιο Ταγιάννη, όπως επίσης, που είναι επίσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά με την ιδιότητά του αυτή μας επισκέφτεται ο κύριος ε, Ταγιάννη. Έχει πολύ σημαντικά πράγματα να μας παρουσιάσει. Έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα ε, για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα. Έχουμε και τον κύριο Ντάλι μετά, Οπότε το πρόγραμμά μας είναι να ακούσουμε το πρόγραμμα εργασίας του για το συγκεκριμένο θέμα, να κάνετε και εσείς ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ε, να κάνετε ερωτήσεις και σχόλια, αλλά στοχευμένα. Συνεπώς, θα ήθελα να καλέσω είτε τους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων είτε τους συντονιστές να κάνουν κάποιες ε, εισαγωγικέ παρατηρήσεις και μετά θα ακούσουμε και κάποια, ε, κάποιες ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας για σήμερα το απόγευμα. Αντώνιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και σου δίνω το λόγο να μας πεις περισσότερα για το πρόγραμμα εργασίας σου. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. αλλά ήμουνα με τους 27 υπουργούς του για να συζητήσουμε για ένα ψήφισμα, μία απόφαση σε σχέση με τον τομέα αυτό που δεν ήταν καθόλου ε, εύκολο. Τώρα θα σας μιλήσω στα Ιταλικά. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι σε αυτήν την αίθουσα η οποία είναι νέα για εμένα αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι να σας μιλήσω στην Επιτροπή σας, στην ΙΜΚΟ, όπου ξαναβρίσκω αρκετούς συναδέλφους που τα προηγούμενα χρόνια είχαν συνεργαστεί μαζί μου στο κοινοβούλιο αυτό. και στα πλαίσια ενός καλώς διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις εργασίες, το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε το Μάρτιο στα πλαίσια του τομέα που είναι της δικής μου αρμοδιότητας. Δηλαδή το πρόγραμμα πρωτοβουλειών που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική που ορίζει το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Οι σχέσεις μου με το Κοινοβούλιο δεν είναι καθόλου τυπικές. 14 χρόνια ήμουν μέλος αυτού του σώματος και γι' αυτό είναι απόλυτα λογικό να έχω μια συνεχή επαφή και άτυπη επαφή με τους ε, βουλευτές, με τους ευρωβουλευτές. Γι' αυτό είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε. Και θα είμαι στη διάθεσή σας ε, κάθε φορά που το επιθυμείτε. Δεν απέχουμε και πολύ. Ε, δηλαδή τα κτίρια τα οποία μας στεγάζουν μία νέα βιομηχανική πολιτική είναι κάτι το πολύ σημαντικό και είναι στο επίκεντρο των στόχων της Ευρώπης 2020. Για να εγκριθεί στα πλαίσια της έγκρισης αυτής της ε, νέας βιομηχανικής πολιτικής, ο πρόεδρος Μπαρόζο αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα επιτρόπων που ασχολούνται με την βιομηχανική πολιτική και εγώ θα συντονίσω τις δραστηριότητες αυτής της ομάδας που θα συζητήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα ενταχθούν στην ανακοίνωση με βάση τα ελλείμματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στους διάφορους τομείς. Έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμευση να ορίσουμε μια νέα και δυναμική βιομηχανική βάση, βάση εργασίας. Θα πρέπει να είναι οριζόντια πολιτική, ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη, αναδιαρθρωμένη, καινοτόμα, να οθεί στη δημιουργικότητα, να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, να, είναι, να αποτελεί μια συνολική στρατηγική και να είναι ολοκληρωμένη. Οι πολιτικές μας θα πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Και βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή διαχείριση, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνουν και τα κατάλληλα, να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα αναδιάρθρωσης στο βιομηχανικό τομέα θα πρέπει να ορίσουμε και ένα σύστημα κανόνων για την προσπελασιμότητα από τους οικονομικούς φορείς. Έχουμε κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός, όμως δεν έχουμε φτάσει σε μία συντονισμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, όπως θα επιθυμούσαμε. Στον τομέα του αυτοκινήτου θα πρέπει ε, να επαναδημιουργήσουμε αυτό το τομέα και να προωθήσουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή που προώθησε η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των καθαρών οχημάτων. Και θα σας παρουσιάσω την ανακοίνωση αυτή, διότι ξέρω ότι ο πρόεδρος Χάρμπορ προσδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα. Πρόκειται για δύο πυλώνες. Καταρχήν, η βελτίωση των ε, παραδοσιακών κινητήρων και η προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων, των υβριδιακών, των οχημάτων που χρησιμοποιούν ε, υδρογόνο ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Γι' αυτό προτείνουμε να έχουμε μία προσέγγιση ευρύτερη και ουδέτερη τεχνολογικά. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ηλεκτρικά οχήματα και να προωθήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα όμως θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε υδρογόνο, φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα και άλλες παρεμφερείς λύσεις μέσα στα πλαίσια των παραδοσιακών κινητήρων. Μιλάμε για 40 συγκεκριμένες δράσεις με στόχο κατευθυντήριες γραμμές και καινοτομίες στη χρήση τεχνολογιών, βιώσιμων τεχνολογιών, να ορίσουμε στόχους για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2011 και να ορίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και όσον αφορά το, τα ηλεκτρικά οχήματα, θα θέλαμε να είναι σίγουρα σε σχέση με την χρήση τους και σε σχέση με τα παραδοσιακά. Θα πρέπει να γίνεται επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ορίσουμε σημεία επαναφόρτισης, δημόσια σημεία επαναφόρτισης. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε στον τομέα των πιστώσεων υποχρεώσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μιλώντας για αηφόρο και ευφύ ανάπτυξη, θα πρέπει να προωθήσουμε την γενικότερη στρατηγική Ευρώπη 2020 και να μιλήσουμε με την Ισπανική Προεδρία. Για αυτή τη στρατηγική επίσης θα ε, ορίσουμε τη, μια νέα επιτροπή ε, σε επίπεδο CARS 21, διότι οι αξιωματούχοι αυτοί θα είναι σε θέση να ορίσουν μια κοινή πλατφόρμα δράσης. Ε, επίσης, θα πρέπει να προβούμε σε τυποποίησεις. Το... Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ένα από τα πολλαπλά παραδείγματα όπου βλέπουμε τις δυνατότητες τυποποίησης και σε ε, θελούσια βάση σε σχέση με την πρόσβαση στις αγορές. Γι' αυτό θα παρουσιάσω το φθινόπωρο ένα φιλόδοξο πακέτο για την τυποποίηση όπου θα ενέχονται πολλές νομοθετικές πράξεις μαζί με μία ανακοίνωση έτσι ώστε η ευρωπαϊκή τυποποίηση κληρωμένη και αποδυτική. Ε, επειδή είμαι πεπισμένος ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ε, σύγχρονη πολιτική προτύπων, θα πρέπει η πολιτική αυτή να εξαχθεί και, σε εξοκινητικές χώρες και ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες. Οι υπηρεσίες μου αξιολογούν τις επιπτώσεις ε, αυτής της μελέτης, γίνεται δηλαδή μια μελέτη αντικτύπου και στις η 21 Μαΐου θα λήξει αυτή η διαδικασία διαβούλευσης online, η οποία άρχισε στις 23 Μαρτίου. Θα πρέπει επίσης να αρκεστούμε στη δική σας ε, πρόταση πρωτοβουλίας για να εμπλουτίσουμε αυτούς τους συσχετισμούς. Μία ε, βασική προτεραιότητα για εμένα αποτελεί και η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Χαίρομαι, διότι ο πρόεδρος Μπαρόζο ανέθεσε στο Μάριο Μόντι την παρουσίαση μέχρι το τέλος του μηνός, δηλαδή μέχρι τις αρχές Μαΐου, μία έκθεση για να βοηθήσουμε την εσωτερική αγορά να υλοποιήσει όλους τους στόχους της. Η ανάκαμψη της αγοράς, θα πρέπει να μιλάμε για ενιαία αγορά πλέον, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μίας αηφόρου ανάπτυξης και μίας στεναρής και ρωμαλαίας ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω λοιπόν ότι οι προτάσεις σας δυνάμει της έκθεσης Γκρές μας οδηγούν σε μια πλέον ολιστική προσέγγιση για μια στρατηγική περί εσωτερικής αγοράς όπου ο πολίτης κατέχει το, το επίκεντρο αυτής της πολιτικής. Είμαι πεπισμένος ότι μαζί με τον συνάδελφο Μισελ Μπαρνιέ θα συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια της νέας ομάδας επιτρόπων που ασχολούνται με θέματα εσωτερικής αγοράς όπως αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο και που συνδονίζει ο συνάδελφος Μπαρνιέ. Και αυτό για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Άρα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα εμπορεύματα που ε, εγκρίθηκε το 2008 μας δίνει συγκεκριμένες πρωταρχικές απαντήσεις για την εποπτεία της αγοράς για τον έλεγχο και για τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Με αυτή την πολιτική ελέγχου των προϊόντων η Επιτροπή θα ήθελε να ενισχύσει την εικόνα ποιότητας και λογοδοσίας του σήματος ΕΚ. Έτσι θα μπορούν οι πολίτες να αγοράζουν προϊόντα ε, ασφαλή προϊόντα οπουδήποτε στην Ευρώπη. Για να επεξηγήσουμε αυτό το σήμα και μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και εμπορευμάτων, εδώ και μερικές μέρες έχουμε ξεκινήσει με μια ευρωπαϊκή εκστρατεία ε, πληροφόρησης για το σήμα CE. Θα λήξει το 2011, κατά τα τέλη του 2011, και έχει ως στόχο της ΜΜΕ. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται δυναμικά σε αυτή τη διαδικασία ως προς την εξέλιξη δηλαδή της εκστρατείας. Ε, ως προς τις μελλοντικές προτεραιότητες θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες απλούστευσης και υπάρχει μία πρόταση που αφορά τους ε, ελκυστήρες και η πρόταση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το ε, καλοκαίρι. Βλέπω ότι ο κύριος Σφάπ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, έτσι δείχνει. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τον αριθμό ε, νομοθετικών πράξεων σε σχέση με παρόμοια κείμενα τα οποία έχει καταρτήσει ο ΩΣΑ και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σε σχέση ε, τώρα με τα οχήματα τύπου L, δηλαδή ε, τρίκυκλα και τετράκυκλα, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για την απλούστευση της κατηγορίας L. Αυτή η αναθεώρηση θα προβλέψει, θα προσπαθήσει να προβλέψει και να, μάλλον να οδηγήσει στην πρόληψη ατυχημάτων σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και μια πρόταση οδηγίας σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής, ιδιαίτερα σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών. Και στο τέλος του 2010 θα υποβάλω μία οδηγία σε σχέση με τον εξοπλισμό ραδιοσυχνοτήτων στα διάφορα τερματικά τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για την οδηγία RTTE και θα σας μιλήσω για τις πρόοδους που έχουν επιτελεστεί σε αυτό το τομέα. Στα πλαίσια του πακέτου περί εμπορευμάτων ορίζουμε ε, μία ε, νέα νομοθεσία δυνάμει της απόφασης 768 κάθετος 2008 έτσι ώστε να ενισχύσουμε την διαδικασία συμμόρφωσης αυτών των προϊόντων ή εμπορευμάτων. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σήμερα επιτάπητος ιδιαίτερα ως προς την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών που έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια του Small Business Act γιατί από αυτήν ε, εξαρτάται το μέλλον των ΜΜΕ. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή σας σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ενέκρινε την έκθεση της κυρίας Βάιλερ με βάση ορισμένου συμβιβασμού τους οποίους φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ μας στο Στρασβούργο. Το, την ψηφίσατε ή θα την ψηφίσατε. Α, την ψηφίσατε. Καλά το είπα, λέει ο Επίτροπος. Η κυρία Βάιλερ θα σας πει αργότερα, θα σας μιλήσει γι' αυτό, λέει ο κύριος Χάρμπορ. Ε, έχει παρέλθει ένας χρόνος από την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση αυτής της πρώτης επιτροπής και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όλους διότι το συζήτησα με εσάς, καταβάλλονται πολλές και μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε, για να εγκριθεί μάλλον από το Κοινοβούλιο ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να είναι αποδεκτό, να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο, έτσι ώστε σε πρώτη ανάγνωση να έχουμε ε, διατάξεις και προδιαγραφές ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες και τις ΜΜΕ που αποτελούν την, τον ακρογωνιαίο λίθο της ε, οικονομίας μας. Μίλησα με πολλούς από εσά και είμαι πεπισμένος ότι ορισμένες από τις πρωταρχικές σας ιδέες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε να προωθήσουμε έναν πραγματικά επικοδομητικό διάλογο με το Συμβούλιο και για να προβάλλουμε τις απαιτήσει και του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές το, ε, το βέλτιστο είναι εχθρός του καλού. Γι' αυτό θα πρέπει ε, αντιστρέφοντας τα πράγματα, να μην χάσουμε άλλον ένα χρόνο. Εμείς οι Ιταλοί είμαστε πολύ καλοί σε συμβιβασμούς, όπως ξέρετε, ακόμα και αν είναι επώδυνοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρακαλέσω να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια ως ΙΜΚΟ και με άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να ικανοποιεί όλους. Στο τέλος πάντα βρίσκεται μια λύση θετική για όλους. Έτσι ώστε να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες που αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις ότι τα καταφέραμε. Βεβαίως όλα μπορούν να βελτιωθούν, αλλά τουλάχιστον τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να συντονιστούν για να δώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά ήθελα να σας πω με λίγα λόγια. Είμαι στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις και είμαι στη διάθεσή σας γενικότερα. Όποτε θέλετε να συναντηθούμε για να σας διευκρινίσω ορισμένα σημεία του προγράμματός μας. Μπορούμε να βρισκόμαστε και στο Στρασβούργο όποτε θέλετε. Σας για ε, την καθυστέρηση που δεν οφειλόταν σε εμένα αλλά στο πρόγραμμα εργασίας. Uh, well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Τα περισσότερα προγράμματα που εγγράψατε στο πρόγραμμά σας και για το οποία έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ακριβώς τον σημαντικότατο ρόλο που καλείστε να παίξετε στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή μας ε, είχε πολύ απογοητευτεί που δεν είχε περισσότερες ε, ευκαιρίες να σας κάνει ερωτήσεις ε, κατά την ακρόασή σας. Εντάξει είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας είναι περισσότερο αρμόδια από μας, όμως ε, όλα αυτά που μας είπατε δείχνουν ακριβώς πόσο μεγάλο είναι και το δικό μας μερίδιο και πόσο σημαντική είναι η δουλειά σας και για την εσωτερική αγορά. Υπήρξαν ορισμένα, αναφέρατε, ορισμένα μεγάλα προγράμματα όχι μόνο ο κύριος Φαμπ, αλλά και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ελκυστήρες. Οπότε, ε, Χαίρομαι που τους έχετε συμπεριλάβει. Εμείς έχουμε ρεκόρ στην αντιμετώπιση πολύ τεχνικών εκθέσεων, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές ε, τις ε, παραεπεξεργαζόμαστε από απόψε ως διατύπωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να καταλήξουμε τελικά και σε μια καλή πρόταση, ενδεχομένως και τέλεια, όπως είπατε κι εσείς. Μέχρι τις 4.30 η ώρα θα είναι μαζί μας ε, ο κύριος ε, ε, Ταγιάννη και ζητήσαμε και από τον Επίτροπο Ντάλι να έρθει λίγο αργότερα επειδή καθυστερήσαμε. Να περάσουμε στις ερωτήσεις τώρα. Δεν ξέρω, ο κύριος Φάμπη κυρία Κόμη. Α, κυρία Κόμη θα πάρει το λόγο. Μετά η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Μπουζόη είναι εδώ, η κυρία Ρούλε, ο κύριος Κότσουσνικ, είναι και ο εισηγητή για τα πρότυπα, την έκθεση πρωτοβουλίας μας, επομένως θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο κύριος De Jong, η κυρία Βάιλερ, η κυρία Στήλερ. Θέλει κανείς άλλος ε, να ε, συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Βάλιρ θα σας ενημερώσει και για τη σημερινή ψηφοφορία. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο λίγο νωρίτερα στην κυρία Βάιλερ. Ας αρχίσουμε με την κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την σαφή σας εισήγηση. Μιλήσατε για συγκεκριμένα θέματα και προτάσεις. Ορισμένες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και άλλες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Χάρβο και τον κύριο Σβάμπ για αυτό το οργανισμό για τους ελκυστήρες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι, όχι, εντάξει, όχι και στις παραλίες, τέλος πάντων. Ε, με συγχωρείτε, ήταν μια καθαρά Ιταλική παρέμβαση αυτή. Σε σχέση με το θέμα που αφορά τις ΜΜΕ, θεωρούμε ότι η Επιτροπή μας ε, Εσωτερικής Αγοράς θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου. Και αυτό που έχει σημασία είναι η απλούστευση των διαδικασιών, όπως είδαμε σήμερα το πρωί για την ανάκαμψη της οικονομίας, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, την οποία θα πρέπει να ανακτήσουμε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Άρα τάσομαι υπέρ ε, της πρόθεσης της Επιτροπής να προβάλλει 46 προτάσεις που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια. Το άλλο θέμα αφορά την ψηφιακή ατζέντα και το διαδίκτυο. Ίσως στα πλαίσια μιας αγοράς θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια ε, εναρμόνιση και συνοχή με στοιχεία που, όπου δεν υπάρχουν φυσικά προσκόμματα. Το διαδίκτυο είναι ένα ε, σημαντικό μέσο και για τους νέους. Το ίδιο θα πρέπει να αφορά το ευρυζωνικό σύστημα έτσι ώστε να έχουμε ομοιογενή χαρακτήρα ανάπτυξης και δεν θα ήθελα αυτή η αυτές οι δυσκολίες να συνεχίσουν να υπάρχουν για τις ΜΜΕ έτσι ώστε να μην υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν δυσκολίες ως προς την κύρωση των διαφόρων κανονιστικών πλαισίων, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τις κοινοτικές πράξεις στο εσωτερικό της ενίας αγοράς. Όπως ε, γνωρίζετε, και επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής είναι πολύ δύσκολη μερικές φορές η επικοινωνία in situ, δηλαδή να δείξουμε στους πολίτες τι εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι οδηγίες και οι κανονισμοί έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με την οικονομική κρίση και να την ε, αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και για το ενδιαφέρον σας για τις ΜΜΕ. Um, να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Βάιλερ, γιατί ξέρω ότι πρέπει και να φύγετε. Θα ενδιαφέρε πολύ την Κομισιόν να ακούσει τη δική σας ανάλυση για το προ... από το πρωινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις πληρωμές. Ναι, Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάω στον ε, γιατρό, οπότε ευχαριστώ που με, που με επιτρέπετε να αναφέρω σήμερα τι έγινε το πρωί. Εμείς οι προβουλευτές νομίζω κάναμε το καθήκον μας όπως έπρεπε. Είχαμε 20 τελείως διαφορετικές θέσεις και καταλήξαμε σε μία. Βρήκαμε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ε, βρήκαμε μια λύση η οποία μπορούσε να γίνει ανοιχτή από όλους από 20 διαφορετικές απόψεις σκεφτείτε. Οπότε τώρα σε εσά είναι το μπαλάκι. Και στις συζητήσεις που θα κάνετε με το Συμβούλιο, από τις 27 θέσεις που θα υπάρξουν στο Συμβούλιο, να βρείτε μια ανεκτή θέση. Εγώ αν θέλετε από Δευτέρα 8 το πρωί θα είμαι στη διάθεσή σας για συζητήσεις. Νομίζω ότι τότε συνεδριάζει και η πρώτη ομάδα εργασία στο Συμβούλιο. Οπότε, τώρα βρίσκεται το μπαλάκι στο γήπεδο του ε, Συμβουλίου. Αν το Συμβούλιο είναι τελείω αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό που ψηφίσαμε εμεί σήμερα το πρωί, τότε μετά το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε. Εμεί είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι κάθε ομάδα είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Κάθε ομάδα έπρεπε να πλησιάσει λίγο την επόμενη, την διπλανή τη. Όλοι καταφέραμε κάτι που να μπορούμε να το δεχτούμε. Οπότε, νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Και επίση θα με ενδιαφέρε πολύ και ο επίτροπο Μπαρνιέ το είπε σήμερα το πρωί, πόσο, σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η απόφαση αυτή για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ειδικά στην ε, περίοδο χρηματοπιστωτικής και οικονομική κρίση που περνούμε, με την, ε, θέλουν δυνατότητες ε, πίστοση, θέλουν θέλουν να έχουν δυνατότητα ε, ρευστότητας. οπότε πραγματικά αυτό είναι ένα ορόσημο. Εσεί τώρα έχετε το παιχνίδι στα χέρια σα. Ε, την απάντησή σα δυστυχώς δεν θα την ακούσω, αλλά θα ενημερωθώ για το τι θα πείτε. Εγώ είχα ε, μπλακεί και στο ε, πακέτο για τα προϊόντα, για τα αγαθά και είχαμε πει τότε ότι περιμένουμε από την Κομισιόν μία ουσιαστική νέα ιδέα για την, ε, για την επισήμανση κτλ. Και τότε δεν είπαμε ότι θα παρατήσουμε την εθνική επισήμανση πριν βρούμε την ευρωπαϊκή κατάλληλη επισήμανση, αλλά και αυτό έχει περάσει καιρός που έγινε. Ε, μετά ήρθε η Νέα Επιτροπή, παρ' όλα αυτά όμως έγιναν οι εκλογέ ήρθε η Νέα Επιτροπή, παρόλα αυτά η Κομισιόν θεωρώ ότι πρέπει να υποβάλει μια νέα επισήμανση, ένα νέο σήμα για ποιότητα για την για τη βιομηχανία, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει προχωρήσει ω προ αυτό. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε στου συναδέλφου μου πόσο συγκεκριμένα είναι τα σχέδια που έχετε για αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Βάιλερ. Την κυρία Γκέπχαρτ τώρα να ακούσουμε και μετά τον κύριο Βουζόη Εντάξει. Αν πρέπει να φύγετε ε, καλύτερα να απαντήσει τώρα ο επίτροπο οπότε να ακούστε και την απάντησή του και μετά ακούμε τις άλλε δύο ε, παρεμβάσεις της κυρίας Γκέφχαρτ και του κυρίου Μπουζόη. Ε, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω προς την κυρία ε, Κόμη. Μίλησε για το θέμα της απλούστευσης του γραφειοκρατικού και διοικητικού φόρτου. Χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, το Διευθυντήριο μάλλον των Επιτρόπων, ενέκρινε την πρόταση απλούστευσης του 7ου προγράμματος δράσης στον τομέα της έρευνας και κινείται, μπορώ να πω, προς αυτή την κατεύθυνση. Κινούμαστε προς την απλούστευση των ε, κανονισμών που προϋπάρχουν και εκεί όπου δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις διατάξεις προσπαθούμε να αλλάξουμε πρότυπο. Και τα στοιχεία που τονίσατε για την ηλεκτρονική ατζέντα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Μπορώ να σας ε, πω ότι θα μιλήσω με την κυρία Κρούς για αυτό το θέμα διότι είναι συνυπεύθυνη, συναρμόδια και θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση που εσείς ζητήσατε. Σε σχέση ε, με την κυρία Βάιλερ, μιλήσαμε με την κυρία Βάιλερ και στο Στρασβούργο. Convinto che un accordo si possa trovare, già come ho eh, parlato. Και επειδή μίλησα με πολλούς ε, βουλευτές ήδη και με εκπροσώπους της Ισπανικής Προεδρίας, έκρινα ότι θα πρέπει να γίνει μια διαμεσολάβηση ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και κρατών μελών για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές με απασχολεί περισσότερο ε, μία ε, ψηφοφορία πριν από το καλοκαίρι και να μην φτάσουμε στην ε, δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή να μην ολιστήσουμε προς τη δεύτερη ανάγνωση, διότι εάν δεν φτάσουμε σε μία συμφωνία θα χάσουμε ένα χρόνο. Και δεν μπορούν να βρίσκονται σε στάση αναμονής ΜΜΕ και οι πολίτες στο μεταξύ. Βεβαίως το Κοινοβούλιο έχει τη θέση του και εμένει σε αυτήν. Ε, είναι και ένα θέμα χρονισμού γενικά. Ξέρουμε που αναφερόμαστε και η μεν και η δε. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία θετική επίλυση. Θα το ξανασυζητήσω με την Ισπανική Προεδρία και με ορισμένα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να πω ότι είμαι απόλυτα αισιόδοξο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πώς, για να σας το πω έτσι. Θα προσπαθήσω να καταστήσω σαφές και στα κράτη-μέλη ότι οφείλουν να λάβουν μία απόφαση σχετικά έγκαιρα. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί και εσείς θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία διαμεσολάβησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Σε σχέση με το πακέτο το, για τα εμπορεύματα και το κοινοτικό σήμα, ακόμα δεν ε, φτάσαμε σε μια τέτοια επίλυση. Δεν φτάσαμε σε ένα σήμα ποιότητας. Ίσως δεν ορίμασαν οι για να φτάσουμε σε ένα σήμα ποιότητας. Εγώ δεν αντιτάσσομαι σε κάτι τέτοιο βεβαίως, αλλά νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να ε, καταστεί γνωστό το σήμα CE πριν μιλήσουμε για ένα νέο ποιοτικό σήμα στην αγορά το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, αλλά δεν αντιτάσσομαι καταρχήν. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να τεθεί σε ισχύ, να γίνει κατανοητό το σήμα CE και μετά να μιλήσουμε για ένα νέο ε, ευρωπαϊκό ποιοτικό σήμα. Ε, ωραία, ευχαριστούμε. Χαίρομαι που απαντήσατε και στην κυρία Βάιλερ. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Γκέφχαρτ τον κύριο Μπουζόη και την κυρία Ρούλε. Να σας θυμίσω ότι μέχρι τις 4.30 τον έχουμε τον Επίτροπο εδώ. Οπότε να είσαστε συνεκτικοί. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που άκουσα την απάντηση πριν μιλήσω. Γιατί μπορώ να απαντήσω και στην, σε αυτά όσα είπε ο κύριος ε, Επίτροπος. Πραγματικά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη ε, δεν ικανοποιήθηκα καθόλου από την απάντηση που δώσατε στα δύο σημεία της κυρίας ε, Βάιλερ. Είπαμε για κάποιες αναβολές για τις πληρωμές. Η κυρία Βάιλερ είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση σε πρώτη, ε, σε πρώτη ανάγνωση αν το Συμβούλιο δεν συμφωνήσει με αυτό που έχουμε ε, προτείνει εμεί. Και ένα είναι απόλυτα σαφέ, κύριε Επίτροπε. Εδώ ψήφισε μια επιτροπή, όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε οι δυνατότητες ε, χειρισμών είναι πολύ περιορισμένες. Αν το Συμβούλιο δεν έχει ήδη άποψη, τότε δεν έχει κανένα λόγο να περιμένουμε και να λέμε και να ξαναλέμε τα ίδια. Ε, καλύτερα θα ήταν και πιο διαφανή και από πολιτικής άποψης έναντι των πολιτών μας να, κα, να καταλήξουμε, να κάνουμε την πρώτη ανάγνωση μάλλον στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβει άμεσα τη δική του απόφαση. Και ίσως να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πραγματικά το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Συμβουλίου να μας πούν τι θέλουν και σε ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν και πόσο είσαστε εσείς διατεθειμένοι να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι ε, εμείς θα μετακινηθούμε. Ε, ε πρέπει να ξέρουμε εσείς τι θέλετε καταρχήν. Αυτό είναι σαφέ. Πέρα από αυτό. Και ήσασταν και εσεί ε, Ευρω... Ε, Ευρωβουλευτή, κύριε Ταγιάννη, και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για του Ευρωβουλευτέ να διατηρήσουν τα δικαιώματά του. Και τα ε, δικαιώματά μα είναι η διαφάνεια των αποφάσεων έναντι των πολιτών μα. Και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή εκπροσωπούνται όλε οι ομάδε. Αλλά όχι όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε ποτέ δεν έχουμε απόλυτη 100% ασφάλεια ότι σε μια ολομέλεια θα, θα υιοθετηθεί αυτό που υιοθετήθηκε ή που ψηφίστηκε σε μια επιτροπή. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας στις διαπραγματεύσεις μας. Γι' αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό από μένα σε αυτό που απαντήσατε στην κυρία Βάιλερ. Δεύτερο σημείο. Ε, τα σήματα ΣΥΗ. Ο προηγούμενος επίτροπος, ο κύριος Φερχόιγεν, ο προκάτοχός σας είχε πει σαφώς ότι οι προσδοκίες που είχε η Κομισιόν και που διευρύνθηκαν και ο τρόπος που θα προχωρούσε είναι για την εγκατάσταση ενός ευρωπαϊκού σήματος σε σχέση με τα εθνικά, αυτό δεν τίθεται, σε, ε, δεν τίθεται καθόλου ως θέμα στο Κοινοβούλιο, γιατί το δεν είναι το σήμα ΣΥΙ, δεν είναι σήμα ασφάλειας. Θα μπορέσει να είναι σήμα ασφάλειας εάν εξελιχθεί έτσι ώστε να αποτελεί όντως σήμα ασφάλειας. Και αυτό όχι μέσω εθελούσιων εξετάσεων, τεστ από, τα, από τις επιχειρήσεις. Από τρίτους και ανεξάρτητους πρέπει να γίνει η ανάλυση αυτή. Πρέπει λοιπόν να, καταρχήν να χρησιμοποιήσουμε τα σήματα ασφαλείας που έχουμε σε εθνικό επίπεδο και που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη και τα οποία εμπιστεύονται και οι πολίτες μας. Και το ερώτημα Τη κυρία Βάλερ ήταν αυτό. Εσεί είσαστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε προ αυτή την άγουσα. Η, απόφαση, η απάντηση ήταν να θα δούμε και περιμένετε λίγο να το κοιτάξουμε. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για μένα, λυπάμαι. Πρέπει να μου πείτε τι ακριβώ προτίθεται να κάνει η Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα. Και μάλιστα γρήγορα πρέπει να κάνει ό,τι είναι να κάνει για να μπορέσουμε να λύσουμε τέλο πάντων αυτά τα θέματα τη ασφάλεια. Κύριε Μπουζόη και μετά η κυρία Ρούλε, Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν ε, μπορώ να μιλήσω Ιταλικά, όμως θα μιλήσω τη γλώσσα που είναι πολύ κοντά στα Ιταλικά, τα Ρουμανικά που είναι και η γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επιτρόπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ε, παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή αυτά που μας είπατε και βλέπω ότι μα μιλάτε για συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Οικονομία. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην εσωτερική αγορά, συνεπώ και είμαι πεπισμένο ότι μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά χωρί εμπόδια, με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και παροχή υπηρεσιών θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μια ε, βιομηχανία χωρίς ε, διοικητικά εμπόδια, χωρί πολλή γραφειοκρατία, κάτι που σημαίνει ανταγωνιστικότητα σε διεθνέ επίπεδο και ανταγωνιστικότητα ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα. Είδα ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν άμεσα με τα θέματα που είναι επίκαιρα και στη δική μας Επιτροπή. Είπατε ότι έχετε σκοπό να παρουσιάσετε μια αναθεώρηση του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις, του Small Business Act και είπατε κι εσείς ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι βασική προτεραιότητα για σας. Όσον αφορά στη συζήτηση για τις καθυστερημένες ε, πληρωμές, Πρέπει να σας πω ότι η εκδοχή που ψηφίστηκε σήμερα στην Επιτροπή μας είναι μια πραγματική βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές του κειμένου. Είναι γεγονός ότι το μπαλάκι τώρα είναι στη μεριά του Συμβουλίου. Αλλά δεν είναι παγίδα αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας, να σας καθησυχάσω. Δεν θέλουμε καθόλου να χρησιμοποιήσουμε την ανωτερότητά μας. Απλώς είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο ε, μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, αλλά είναι και κάτι το οποίο μπορεί κάλλιστα να το δεχθούν και τα κράτη-μέλη. Είδα επίσης ότι έχετε σκοπό να παρουσιάσετε μια ανακοίνωση σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα, ενό τομέα ο οποίος κατά τη διάρκεια τη ε, οικονομική κρίση επηρεάστηκε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα έχετε σκοπό να αναλάβετε συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης για το συγκεκριμένο τομέα κατά την ε, επερχόμενη περίοδο, γιατί χωρίς συντονισμένη στρατηγική στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένη τη συγκυρία τη οικονομική, δεδομένη τη κρίση, δεδομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζει ο τομέα σε πολλά κράτη-μέλη και κυρίω ε, στα κράτη-μέλη που αναπτύσσονται, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ο τομέας αυτός ε, να ξεπεράσει την ε, οικονομική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος, η κυρία Ρουλέ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Γκέφχαρτ και θα το υπογραμμίσω κι εγώ. Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που είπε. Σήμερα ψηφίσαμε στην Επιτροπή επί σημαντικών ε, συμβιβασμών. Οι διαπραγματεύσει όμως θα ξεκινήσουν όταν θα έχουμε μια κανονική πρώτη ανάγνωση. Πιο πριν δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε για το αποτέλεσμά μας. Αν το Συμβούλιο συμφωνήσει ένα προ ένα, εντάξει, δεν, έχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα, κλείνουμε και στην πρώτη ανάγνωση κατευθείαν. Αλλά ξέρετε ότι έχει, έχει αλλάξει αρκετά με τη δική μα σημερινή ψηφοφορία η πρόταση της Κομισιόν. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μιλούμε για νέους συμβιβασμού. Καταρχήν πρέπει να δούμε αν συμφωνεί το Συμβούλιο μαζί μα Και να τονίσω και κάτι άλλο. Αυτή η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και οι διαπραγματεύσει πίσω από κλειστέ πόρτες δεν είναι πολύ δημοκρατικέ πρέπει να σα πω. Και δίνουν πολύ περιθώριο λιγμό στην Κομισιόν. Και, και εμεί ε, δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται στο Συμβούλιο με τι ε, ε διαπραγματεύσει. Οπότε, επί τη βάση αυτή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τέτοιου είδου συμβιβασμού. Σα το λέω σαφώ. Και να πω επίση ότι για την οδηγία για τα παιχνίδια τα παιδικά, έχουμε πάντα πολλά προβλήματα στη Γερμανία με τα σήματα. Η Κομισιόν είπε ότι θα κάνει μια έρευνα και θα μας, ενα... θα μας δώσει νέα νούμερα, νέα στατιστικά με πριν το καλοκαίρι. Ελπίζω να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλές αρνητικές εμπειρίες, Είμαστε... έχουμε καεί στον τομέα αυτό. Αλλά το είπατε κι εσεί για το πακέτο για τα αγαθά, είσαστε υπεύθυνο και για τον τομέα τη εποπτεία τη αγορά. Και στον, ε, στην εποπτεία τη αγορά υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα στην, ε, στα κρατημέλη. Και αν μιλούμε τώρα για ευρωπαϊκή σήμανση, για, μαρ, για σήμα ΣΥΗ, πρέπει να μιλούμε για, για εποπτεία τη αγορά. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει αυτό να λειτουργήσει σωστά. Να υπάρχει δηλαδή σωστή χρήση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού σήματο τα κράτη-μέλη ήταν ε, διατεθειμένα μετά το πακέτο για τα αγαθά να επενδύσουν περισσότερο και να κάνουν και κάτι περισσότερο. Αλλά και εσεί πρέπει να δώσετε λίγο χέρι στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εποπτεία τη αγορά. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Μήπω θέλετε, κύριε Επίτροπε, να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά. Μερικά συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Ίσως ε, δεν ήμουν σαφής μιλώντας Ιταλικά όταν σας ε, μίλησα για την πρόταση οδηγίας για την καθυστέρηση των πληρωμών. Δεν ζήτησα από το Κοινοβούλιο να αλλάξει θέση, επουδενή. Απλώς επειδή θέλουμε να απαντήσουμε σε εκατομμύρια ΜΜΕ που δίνουν εργασία σε εκατομμύρια ανθρώπων και επειδή γνωρίζουμε το πρόβλημα, ε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η δανειοληψία και η καταβολή των πληρωμών εγκαίρως, γιατί διαφορετικά ε, πολλοί πολίτες θα χάσουν την εργασία τους. Εγώ μιλώ για ένα κοινωνικό πρόβλημα πρωτίστως κοινωνικό. Γι' αυτό ζητώ από το Κοινοβούλιο να μην παραβιάσει κανέναν κανόνα, να χρησιμοποιήσει όλα του τα προνόμια, γιατί εγώ πάντα μιλούσα πολύ καθαρά. Το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι επιθυμεί. Εγώ λέω απλώς ότι προς συμφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων θα ήταν σκόπιμο να εγκριθεί το κείμενο της πρότασης οδηγίας στην πρώτη ανάγνωση. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει να δεχτεί τις προτάσεις του Συμβουλίου, εάν το Συμβούλιο δεν θέλει να δεχτεί τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, δεν είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Γιατί οι γάμοι γίνονται μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αλλιώ θα χάσουμε ένα χρόνο. Εγώ κάνω μία έκκληση, αλλά έκανα έκκληση όχι μόνο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη δική σας Επιτροπή, έκανα έκκληση και προς το Συμβούλιο. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί για την επίτευξη συμφωνίας. Τα προνόμια σας είναι αυτά που είναι. Ασκείτε πολιτική εσείς θα κρίνετε πώς θα επιτευχθεί μία συμφωνία και πώς θα φτάσετε σε συμβιβασμούς. Γιατί μπορεί να επιτευχθεί ένα συμβιβασμός ακόμα και σε επίπεδο ψηφοφορίας. Αυτό μου δείχνει η 15 ετής μου πείρα. Διότι πολλές φορές για να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους εργαζόμενους, διότι κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών. Δηλαδή, οι ΜΜΕ, αν δεν έχουν έγκαιρες πληρωμές, δεν μπορούν να πληρώσουν και τους υπαλλήλους. Άρα, ζούμε σε μία περίοδο κρίσης, μία άκρος ιδιάζουσα περίοδο. Γι' αυτό έκανα αυτή την έκκληση. Θεωρώ ότι η καθήκον μου είναι να προωθήσω αυτή τη θέση ενώπιον και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έκανε έκκληση και στο Συμβούλιο. Μίλησα με την Ισπανική Προεδρία έτσι ώστε να παρέμβει σε επίπεδο κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορέσει να εξευρεθεί μία λύση το συντομότερο δυνατόν. Δεν θέλω να ε, παραβιάσω το πλαίσιο προνομίων σας. Ως προς το Ευρωπαϊκό Σήμα, γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Σήμα δεν είναι ένα σήμα ασφαλείας. Και σας το λέω με λίγα και φτωχά λόγια. Η Επιτροπή δεν θα δημιουργήσει ένα σημείο ποιότητας τώρα. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σήμα αρκεί. Έχει αρχίσει μία εκστρατεία για να γνωστοποιηθεί το σήμα αυτό στους ε, πολίτες. Θα πρέπει η Επιτροπή να παρέμβει σε επίπεδο κρατών μελών για να υπάρξει πραγματική εποπτεία, όχι μόνο τυπική, όχι μόνο τύπης θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αντιτίθεμαι σε ένα σήμα ποιότητας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Ας προωθήσουμε το ευρωπαϊκό σήμα που δεν είναι ποιοτικό σήμα, αλλά μιλά για την τήρηση των ε, προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Αλλά δεν είναι ε, προϊόν ποιότητας καθαρά. Ως προς τα οικονομικά δεδομένα συμφωνώ. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, παρούσα κρίση χωρίς συντονισμό, χωρίς μια οικονομική πολιτική γιατί δεν θα πρέπει να προβάλλουμε εθνικισμούς και προστατευτισμό. Αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Ίσως επιφανειακά σε κάποιους αρέσουν αυτές οι εθνικές και προστατευτικές προσεγγίσεις, αλλά για όποιον ασχολείται με την εσωτερική αγορά, ε, ο, αυτός οφείλει να καταδικάσει εθνικιστικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για την άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, δηλαδή εσωτερική αγορά και συντονισμένες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα στον κατασκευαστικό τομέα, βλέπω ότι παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μου. Θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι προτίθεμαι να προωθήσω μία μελέτη για να δούμε πώς θα ε, ενισχύσουμε τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά ε, δεν έχουμε ακόμα ορίσει την στρατηγική μας. Είμαι πεπισμένος ότι πριν ορίσουμε τις επιλογές μας, πριν τις προσδιορίσουμε θα πρέπει να προβούμε σε μία μελέτη αντικτύπου, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας στον περιβαλλοντικό τομέα. Είναι πρόωρο να ορίσουμε, να προσδιορίσουμε το πλαίσιο με μία ακριβή πρόταση. Υπάρχει βεβαίως η θέληση αυτή υποστήριξης του τομέα γιατί για ορισμένα ποιοτικά ε, προϊόντα οι αγορές έχουν προσαρμοστεί. Γνωρίζουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας γνωρίζει μεγάλες δυσκολίες όπως στην Ισπανία, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες Γι' αυτό σας είπα ότι η πρόθεσή μου είναι να συνεργαστώ για την ανάκαμψη. Τώρα κινηθήκαμε για τα οχήματα, μετά για την καινοτομία. Έχουμε πολλά στα σκαριά και επειδή είναι ένας ιδιαίτερος τομέας, θα συνεργαστούμε και θα λάβουμε υπόψη όλες σας τις υποδείξεις και γι' αυτό μετά θα κινηθώ και για αυτό το σχέδιο που αφορά τον τομέα κατασκευών. Για να συνεισφέρουμε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε καθυστερήσει. Θα σας πω ποιοι είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Κώσης θέλω επίσης να πάρει το λόγο, για να, γιατί είναι και ο εισηγητής, Ντεγιόν, Μάντες, Σφάμπ, Στήλερ και κυρία Μπίλτς. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας περιορίσω πάρα πολύ στο χρόνο, αλλά δέκα λεπτά μας απομένουν, οπότε ένα λεπτό, δύο λεπτά το πολύ. Θα σας χρονομετρούμε κιόλα για να σας βοηθήσουμε. Κύριε Σκότσισνικ πρώτα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας εκ μέρους της δικής μου ομάδας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ την ε, εφαρμογή του προγράμματος αυτού, γιατί δεν μας μένει πάρα πολύς χρόνος για όλα αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε. Έχουμε επενδύσει τα πάντα και το ζήτημα είναι πώς θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω λοιπόν να σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας. Άκουσα και κάτι που είπατε και που μου άρεσε πάρα πολύ. Ανταγωνιστικότητα. Πολύ μου άρεσε ο όρος αυτός που χρησιμοποιήσατε, γιατί ένας πολιτικός στη δική σας θέση, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση που καταπολεμά την κρίση, πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα. Και ένας από τους όρους της ανταγωνιστικότητας είναι βέβαια και η τυποποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ε, Επιτροπή μας και έχουμε και μία έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Και εγώ ως εισηγητής, μαζί με άλλους εισηγητές, ε, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στι 23 Ιουνίου σε μια ακρόαση για το μέλλον της ευρωπαϊκής Τυποποίηση. και ελπίζω να καταφέρετε να βρείτε λίγο χρόνο για να έρθετε. Ο κύριος Φερχόγγιν, ο προκάτοχός σας, ασχολήθηκε επίσης με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ε, ο κύριος Μπαρόσο, το έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και εκείνος. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς έχουν τα πράγματα τώρα όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δε Ιόγκ. Ehm, eh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι αυτά που μας είπατε πραγματικά συνάδει με όλα αυτά που θέλουμε και εμείς να κάνουμε. Είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε παράπονα από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μας λένε ότι έχουν ε, να αντιμετωπίσουν άχρηστου κανόνες, άχρηστε ε, διαδικασίες. Επομένως υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να απευθύνουμε ως έκκληση προς όλους τους επιτρόπους Υπάρχει μια δυνατότητα να σας γνωστοποιούμε τα παράπονα αυτά και να μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν σε εσά ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Επίση, η εσωτερική αγορά είναι επίση πολύ σημαντική και για τους πολίτες, για όλους τους καταναλωτές. Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά όταν βλέπουμε τι γίνεται με την ηλεκτρονική ατζέντα, για παράδειγμα, και στην κυρία κρούστο θέσαμε το ερώτημα αυτό. Τι γίνεται με το ίντερνετ και κυρίως με τους πιο ηλικιωμένους ε, πολίτες ώστε να έχουν πρόσβαση και εκείνοι. Καινοτομία, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Συγχαρητήρια για αυτά που μας είπατε, αλλά γνωρίζουμε όλοι οι περιόδους ισχνών αγελάδων, προβλήματα στον προϋπολογισμό για όλα τα κράτη-μέλη. Θα, μπορού, θα μπορέσουμε λοιπόν να διαθέσουμε επιπλέον πόρους στην έρευνα, για παράδειγμα, που θα ήταν κάτι το πολύ χρήσιμο. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις καινοτομίε για το διαδίκτυο, για να μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα όλων των επιχειρήσεων, όλων των πολιτών, των καταναλωτών, πώς θα τα ελέγξουμε όλα αυτά και παράλληλα να μην σπαταλούμε και πόρους. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε ταμεία, για παράδειγμα, για την καινοτομία. Αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν γίνεται σπατάλη χρημάτων, ενώ θα τα χρειαστούμε αυτά τα χρήματα σε τομεί πολύ σημαντικούς. Για τις καθυστερημένε πληρωμές τώρα. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα σχέσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όχι, είναι ζήτημα άποψης για ένα συγκεκριμένο θέμα, την οποία έχουμε και θέλουμε να γίνει σεβαστή. Αν σα ενδιαφέρουν λοιπόν τόσο πολύ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα έπρεπε να μην σα διαφεύγει ότι αυτέ οι επιχειρήσει ζήτησαν κανόνε πιο ευέλικτου. Και επίση να πληρώνονται κιόλα. Άρα το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό τη καθυστέρηση των πληρωμών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές και μετά θα δώσω στον Επίτροπο το λόγο να απαντήσει σε, σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί θα έρθει και ο κύριος Ντάλι πολύ, πολύ σύντομα. Μάντερ, Σφαμπ, Στήλερ και Κρότσπιλς. Κύριος Μάντερ. Ευχαριστώ πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα της εσωτερικής αγοράς, από όπου προκύπτουν όλα τα προβλήματα, και τα παράπονα είναι η εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών και ελπίζω ότι κατά τα ερχόμενα έτη θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα με όλ, σε όλον αυτόν δηλαδή τον νομοθετικό μηχανισμό που πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που δεν ισχύει τώρα. Στη δική μου, στην, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μιλήσαμε επίση και για την ευθύνη των ε, ε διευθυντών, ε, των ε, επικεφαλής των επιχειρήσεων για να μην κάνουν κατάχρηση της θέσεώς τους. Να έχουν δηλαδή αστική ευθύνη. Όχι μόνο πρόστιμα να πληρώνουν, που ούτως ή άλλως η επιχείρηση θα τα πληρώσει. Όσον αφορά τώρα την ετικετοθεσία για τα υφάσματα. Ελπίζουμε ότι και εσείς αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσετε να μας υποστηρίξετε στο Συμβούλιο. Εμείς, ως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών, ήμασταν σαφέστατοι. Είπαμε ότι προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι αντικείμενο ενημέρωσης συγκεκριμένης ε, ε, για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα γιατί εκείνα ε, ζητούν τέτοιου είδους πληροφορίες και άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Προς όφελος του καταναλωτή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάντερς. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο Ντάλη και την ομάδα του. Να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας με τον κύριο Ταγιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εγκαίρως. Σφαμπ, Στήλερ και Κρότσελ Πίλκ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Αντώνιο, Εκ μέρους τη ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για τι καθυστερημένες πληρωμές, για το σχετικό πακέτο. Ήταν πραγματικά επικοδομητικές συζητήσει, παρόλο που υπήρχαν κάποια σημεία για τα οποία ήταν διαφορετικέ οι απόψει μα. Σε ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Για το ερώτημα του κυρίου Ροσφόρ για το πώς θα προχωρήσουμε. Ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί. Σωστό είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει μια απόφαση, αλλά και εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να βοηθήσουμε άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό, ανάλογα με το πώς θα πάει η διαδικασία, ακόμη και μετά την ψήφιση στην Ολομέλεια, ε, θα μπορούσαμε ίσως να ε, ζητήσουμε την, ε, από την εισηγήτρια να δράσει άμεσα γιατί πραγματικά ενδιαφερόμαστε, θέλουμε γρήγορα να φτάσουμε σε μια λύση. Ο Επίτροπο για την βιομηχανία είναι αυτός που έχει τα περισσότερα, τους περισσότερους φακέλους που αφορούν τη δική μας Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια αγαστή συνεργασία και για όσα είπατε να επαναλάβω το εξή. Ε, συσκευασίες και παιχνίδια. Ετέθη πρέπει και αυτά να βοηθήσουν ε, ε, και ο τομέας αυτός να βοηθήσει γιατί παρόλα αυτά οι, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πολλές, πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό. Με κάποιο τρόπο λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το τι γίνεται στον τομέα αυτό προς το κοινό και χαίρομαι ε, για τις πρωτοβουλίες που ελπίζω να μα υποβάλει η Κομισιόν ω πακέτο για τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τρία σημεία πολύ σύντομα όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Υπάρχει στη Γλασκόβη η OI Vehicles, ε, η οποία δοκίμασε ένα από τα ηλεκτρονικά της οχήματα πέρσι κατά την προεκλογική εκστρατεία. Και έχω ενθουσιαστεί με την επένδυση που έκαναν στα πρότυπα. Ξέρω τι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώ αυτή η σκοτσέζικη εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην όλη διαδικασία τη ευρύτερη τυποποίηση, όσον αφορά τώρα τον κατασκευαστικό τομέα. Όπω γνωρίζετε, είμαι η συγγήτρια για αυτό το θέμα που έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί για την ώρα τα πράγματα έχουν μείνει στάσιμα. Ελπίζω να επιστρέψει το κείμενο για δεύτερη ανάγνωση το στομότερο δυνατό. Και πάλι για την τυποποίηση. Χαιρετίζω την πρόταση για την ε, τυποποίηση. Τέλη Μαΐου θα πάμε στην Ελβετία για το ζήτημα αυτό της τυποποίησης και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να ορίσουμε τα δικά μας πρότυπα, αλλά να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα. ψηλότερα πρότυπα σημαίνουν καλύτερη προστασία για τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βίλτ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας είναι μία από τις προτεραιότητές σας γιατί φυσικά η ΜΜΕ ο ακρογωνιαίος λήθος της κοινωνίας μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς θα κάνετε για να θέσετε σε εφαρμογή την ε, λεγόμενη smarter legislation. Νομίζω ότι θα πρέπει ότι θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ μια συμφωνία. Αν δεν ξέρω πια να μιλάω Ιταλικά, λέει ο Μιλήτρια. Για να ταχθούμε υπέρ της συμφωνίας με το Συμβούλιο, διότι υπάρχουν ΜΜΕ που αναμένουν απάντηση. Για την τυποποίηση θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα συμπεριληφθεί η πραγματογνωμοσύνη των επιχειρήσεων. Πώς θα ληφθεί υπόψη κατά την διατύπωση της πρότασής σας. διότι υπάρχουν πολλές γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Επίτροπε, αλλά νομίζω ότι θα θέλατε να σχολιάσετε ε, ορισμένα ε, ζητήματα λεπτομερίας που έθιξαν οι συνάδελφοι. Σας δίνω το λόγο. Εγώ δεν έχω μια γραφειοκρατική αντίληψη περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα ό,τι μπορέσω να κάνω για να ε, ε, ελαφρύνω το γραφειοκρατικό φόρτο για τις ΜΜΕ θα το κάνω, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν είμαι υπεύθυνο όπως ήταν ο Επίτροπος Βιομηχανίας για την διοικητική απλούστευση, αλλά ως μέλος της Επιτροπής θα βάλω κάθε προσπάθεια για να επιταχύνω αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν ήμουν επίτροπος μεταφορών επιτάχυνα τη διαδικασία Μάρκο Πόλο. Ε, εν πάση περιπτώσει τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Ως προς το Small Business Act είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κατά τις συζητήσεις Γνωρίζετε ότι προβλέπεται αναθεώρηση το δεύτερο ήμιση του 2010 και αναμένουμε και τη δική σας ανάδραση. Τα δικά σας δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Ε, κύριε Τεγιόγκ, πολλές είναι οι χώρες που εμπλέκονται δεν σημαίνει όμως ότι το Small Business Act θα επιβληθεί ως διαμαγίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ με όποιο τρόπο μπορούμε. Εγώ πάντα επισκέπτομαι τις μικρομεσαίες σε μια χώρα πριν δω τι μέτρα μπορούν να ληφθούν. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα υπέρ των ΜΜΕ δεν θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα. Το θίξαμε με, τον Επίτροπο, με την Επίτροπο Βιομηχανίας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε όμως θα το κάνουμε στα πλαίσια του Small Business Act. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν τις ΜΜΕ με κάθε τρόπο. Και ως προς το Made in, γνωρίζω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξαν επιφυλάξεις εγώ ξέρετε ότι είχα μαζέψει υπογραφές κατά την ε, προηγούμενη θητεία. Δεν μπορώ να απαρνηθώ το παρελθόν μου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εποπτεύσουμε τα προϊόντα μας και την εσωτερική μας αγορά. Δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε το εμπόριο. Θα πρέπει να έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Και το σήμα Made in αποτελεί εποπτεία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας. Μπορεί να μην το συμμερίζονται βέβαια αυτό όλοι. Ως προς την ε, ε, ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας, αυτό σημαίνει και καινοτομία. Καινοτομία σημαίνει τυποποίηση και ούτω καθεξής. Πρόκειται για μια στρατηγική που θα πρέπει να δούμε στο σύνολό της. Όσα ανακύπτουν από τις συζητήσεις αυτές ε, οδηγούν σε μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος και ιδιαίτερα της ΜΜΕ. Εγώ καταβάλω μεγάλες προσπάθειες γιατί θέλω να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι ΜΜΕ. Δεν μπορώ να είμαι αμέτωχος έκανα μία έκκληση γιατί προτίθεμαι να κάνω πολιτική. Ο κύριος Σβάμπ μας ε, υπενθύμησε πολλά πράγματα εγώ ανήκω στη δική του πολιτική ομάδα, αλλά είχαμε διχογνωμίες ή αντιγνωμίες πολλές φορές. Μπάς περιπτώσει το να βρούμε ένα συμβασμό δεν σημαίνει λάθος. Στην πολιτική πάντα πρέπει να βρίσκουμε συμβασμούς. Αν θέλετε να μιλάμε για συμφωνία, συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία συμφωνία και σε επίπεδο τριών θεσμικών οργάνων. Εμείς δεν θέλουμε να επιτύχουμε το 100%. Θα αρκεστούμε σε χαμηλότερη ποσοστή ε, αναλογία. Εγώ μπορώ να κάνω πίσω σε μια αρχική μου θέση. Αν όμως θεωρήσω ότι βρίσκεται μια γενικά καλή λύση, κάνω ένα βήμα προς τα πίσω για να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξαν οι ιδέες μου ή θέλω να προωθήσω ακρεφνείς θέσεις. Κύριε Ντεγιόγκ, μου μιλήσατε για τη συμβατική ελευθερία και τη συμβατική ευθύνη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να εξεύρουμε λύσεις και να κινηθούμε μέσα σε πλαίσια συγκεκριμένου χρονισμού. δεν υπάρχει μία ενιαία και απαράβατη αρχή για όλα. Πρέπει να βρούμε μία καλή ρυθμιστική λύση, διότι δεν θέλουμε ο καθένας ε, να δείξει ότι έχει δίκιο. Θέλουμε να επιτρέψουμε στις ΜΜΕ να μπορέσουν ε, να λάβουν αυτό που επιθυμούν. Το συζητάμε και προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Μακρηγόρησα. Ως προς την τυποποίηση, θα συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Το θεωρώ ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της αγοράς. Εμείς ε, αναθέσαμε το θέμα στον αρμόδιο επίτροπο ως προς την τυποποίηση θεωρούμε ότι μέχρι του χρόνου θα πρέπει να έχουμε μία εναρμόνιση σε σχέση με τα ηλεκτρικά συστήματα επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Θέλουμε λοιπόν ενδείξεις και υποδείξεις από τη βιομηχανία. Εγώ δεν έχω μια γραφειοκρατική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Δέχομαι λοιπόν τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βρούμε ε, καλές και σκόπιμες απαντήσεις. Στόχος μας είναι να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση σε μισό εκατομμύριο πολιτών που προσμένουν μια λύση από μας. Αν δεν μπορώ να το κάνω, κύριε Σφάπ, τότε ε, δυστυχώς θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Δεν σημαίνει ότι εισφάλουν πάντα οι πολίτες. Πολλές φορές έχουν δίκιο, γιατί δεν μπορούμε να τους δώσουμε απαντήσεις. Αν υπάρχουν δόλοι χειρισμοί είναι άλλη υπόθεση. Εμείς όμως προσπαθούμε να δώσουμε τις βέλτιστες δυνατές απαντήσεις μέσα στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε, που ε, ήρθατε σήμερα. Γιατί ο ενθουσιασμός, ο ενθουσιασμός σας και το πάθος σας ε, είναι πραγματικά έκδηλα. Πρόκειται για ζητήματα που θα εξακολουθήσουμε να συζητούμε μαζί σας. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να προοδεύσουμε Ελπίζω να μπορέσετε να έρθετε στην ακρόαση για την τυποποίηση στις 23 Ιουνίου. Ιουνίου. Επίσης περιμένουμε και άλλα ζητήματα να συζητήσουμε όπως τα πράσινα αυτοκίνητα. Είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ενδεχομένως το συζητήσουμε και με τον κύριο Ντάλι. Και υποθέτω ότι η κυρία Στήλερ θα είναι μία από τους πρώτους αποδέκτες ε, του κειμένου που ενδεχομένως να παρουσιάσετε. Θα έρθω, θα έρθω στην ακρόαση, λέει ο κύριος Σταγιάννη. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ντάλι. ladies and um, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, εντατικό το απόγευμά μας σήμερα. Our task has been to squeeze in, uh... Προσπαθούμε να χωρέσουμε τους ε, δύο βασικούς επιτρόπους για να μας μιλήσουν για το πρόγραμμα εργασίας τους. Ο Τζον Ντάλι είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Πρώτη φορά που έρχεστε μετά από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Χαίρομαι λοιπόν που ε, είσαστε εδώ μαζί μας ε, στο πάνελ του Προεδρείου. Ξέρω ότι ήσασταν πάρα πολύ απασχολημένος μόλις γυρίσατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται και με ε, τις δικές μας υποθέσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών. Ξέρω ότι έχετε αρκετά, αρκετές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στο πρόγραμμά σας. Οπότε θα σας δώσω το λόγο και θα καταρτήσουμε και έναν κατάλογο μιλητών. Θα δώσω την προτεραιότητα στους ομιλητές από τις ομάδες, αλλά επειδή παρά ήμασταν επίσημοι, καλό θα ήταν να ακούσουμε κάποιους από τους ομιλητές που βρίσκονται και εδώ στην αίθουσα και μετά να δούμε και τους ε, συντονιστές, γιατί μπορεί να θεωρήσετε ότι ε, σας μειώνουμε συνέχεια το χρόνο ομιλίας. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο χαλαροί αυτή τη φορά. Θα κάνουμε πιο γενικό κατάλογο ομιλητών. Ελπίζω να μπορέσω να δώσω σε όλους σας τη δυνατότητα να μιλήσετε. Τζον, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όπως είπατε, Πρόεδρε, είναι η πρώτη μου συνεδρίαση με την ε, Επιτροπή σας από όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Επιτροπός Υγείας και Πολιτικής για τους καταναλωτές και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Είναι τιμή μου να έχω αυτή τη δυνατότητα σήμερα να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για το πώς σχεδιάζω να αρθώ στο ύψος των υποχρεώσεών μου για την συνεργασία μαζί σας σε ό,τι αφορά τον κοινό στόχο για την υγεία και τους καταναλωτές. Η ε, πολιτική για τους καταναλωτές ε, βρίσκεται πραγματικά στον πυρήνα των προκλήσεων που υπάρχουν για την Ευρώπη ε, του 2020 οι καλώ πληροφορημένοι καταναλωτέ θα αποτελέσουν το κλειδί για την, επιτυχία τη εσωτερική αγορά. Η αλλαγή των ε, συνηθιών των καταναλωτών είναι απαραίτητη αν θέλουμε να έχουμε πιο βιώσιμη οικονομία. Να δημιουργήσουμε, την, ε, να δημιουργήσουμε μια λειτουργό αγορά για του ε, καταναλωτέ, ειδικά του πιο ευαίσθητου, στην καθημερινότητά του, είναι σημαντικό για να επανασυνδεθούμε με του πολίτε. Η σημασία της οριζόντιας διάστασης της πολιτικής για τους καταναλωτές αντικατοπτρίζεται και στο ότι τα θέματα των καταναλωτών αποτελούν τώρα ένα ενσωματωμένο τμήμα των χαρτοφυλακίων πολλών άλλων επιτρόπων παρόλο που αυτό είναι και ε, καλό, θετικό για την, για την ε, αυξανόμενη σημασία της ε, πολιτικής για τους καταναλωτές, αποτελεί και ένα αίτημα για μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Γι' αυτό σχεδιάζω να είμαι σε στενή επαφή και συνεργασία με τους συναδέλφους επιτρόπους και όταν είναι απαραίτητο να κάνουμε και ad συναντήσεις μαζί τους για να συζητούμε θέματα ευρεία στρατηγική ή ειδική στρατηγική που είναι σημαντικέ για, τις, ε, ε, για τους Ευρωπαίους καταναλωτέ. Ήδη έχουμε έναν αριθμό μέσων στη διάθεσή μα που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα για του καταναλωτέ. Το βαθμολόγιο των, ε, για του καταναλωτέ και οι σχετικές μελέτες της αγοράς είναι πολύ καλά παραδείγματα εργαλείων που μπορούν να μα βοηθήσουν να συνεχίσουμε να καταδεικνύουμε και να δείχνουμε πού είναι τα προβλήματα στην αγορά. Έχουμε ε, σημαντικό ποσό ε, δεδομένων ε, για τις, συνθήκες, για τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των καταναλωτών που μπορούν να μας βοηθήσουν να εκπονήσουμε σωστή στρατηγική και να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Εγώ θα ε, χρησιμοποιήσω αυτή την ε, εμπειρογνωμοσύνη των δικτύων των, των, δικτύων, των ε, ενώσεων των καταναλωτών και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τους καταναλωτές. αν θέλουμε όντως να ωφελήσουμε τους καταναλωτές θα πρέπει να αρχίσουμε καταρχήν να τους ακούμε. Καλωσορίζω την πρότασή τη ε, στην έκθεση HED για την ετήσια έκθεση για το πώ ενσωματώνονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Και σα ε, ε, διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω στενά. Συνεργασία μεταξύ του Κολεγίου των Επιτρόπων θα αντικατοπτρίζεται σε οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει σε επίπεδο υπηρεσιών και στην Γενική Διεθνή ΣΑΝΚΟ μαζί με του συναδέλφου, θα, θα εργαστούμε μέσω μια διυπηρεσιακή ομάδα για θέματα καταναλωτών ώστε να συντονιστούμε και να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών ε, ενσωματώνονται στι πολιτικέ τη Κομισιόν. Βέβαια, δεν μπορώ να σα δώσω, να καθορίσω πάντα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τομεακέ πολιτικέ. Ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών δίδονται, στα συμφέροντα των καταναλωτών δίδεται όλη η ε, προσοχή που πρέπει, είναι να προβλέπουμε τι εξελίξει και να επενδύουμε το χρόνο και το χρήμα που χρειάζεται, ώστε να ε, μπορέσουμε να, τα, να ενσωματώσουμε αυτά στις διάφορες αρμοδιότητες των επιτρόπων. Ε, ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ε, παρακολουθούμε με τον ε, Αντιπρόεδρο Ταγιάννη την πρωτοβουλία για τα πράσινα αυτοκίνητα και με, επίσης στην οποία έχει Έχουμε μπει πολύ στενά στην αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τους εγκάρσιους περιορισμούς από τον Αντιπρόεδρο Αλμούνια. Η ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών ε, στι διάφορε πολιτικέ τη Κομισιόν δεν είναι πάντα ε, θέμα του πόσο καλά μπορούμε να, να, να λάβουμε κάποιε πρωτοβουλίε, αλλά πώ μπορούμε να διαχειριστούμε τι ε, προοπτικέ που έχουν οι καταναλωτέ και πώ μπορούμε αυτέ να τι διαχύσουμε και σε άλλου τομεί. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί ε, φάκελοι και εγώ, όπου εγώ έχω μεγάλο περιθώριο κινήσεων και λιγμών και ε, εφόσον πέφτουν στην, εμπίπτουν στη δική μου δικαιοδοσία ή επειδή είτε στα θέματα καταναλωτών είτε στα θέματα ε, υγείας. Ε, ας πούμε η πληροφόρηση των ασθενών και επισήμανση των τροφίμων είναι σημαντικά θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Σας ε, ε λοιπόν ότι έχω την πρόθεση να συνεχίσω αυτές τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Η ευημερία των καταναλωτών είναι το, τελευταίο, βασικό τεστ για την εσωτερική αγορά. Ακόμη και σήμερα, δύο δεκαετίε μετά την δημιουργία τη εσωτερική αγορά, υπάρχουν ε, προσκόμματα τα οποία αποτρέπουν του πολίτε από το να την απολαύσουν στο πλήρε ε, φάσμα τη. Η ατζέντα για την Ευρώπη του 2020 προσπαθεί να ε, απαλείψει αυτά τα προσκόμματα και να βάλει την Ευρώπη στον δρόμο τη έξυπνη, βιώσιμη και συνολική ανάπτυξη. Όταν συναντήθηκα με τον κύριο Μόντι για την προετοιμασία αυτή τη έκθεση, ε, είπα ότι το να δώσουμε ένα νέο κίνητρο στην εσωτερική αγορά και να συνδέσουμε του Ευρωπαίου ε, με μια νέα δυναμική ήταν η μόνη δυνατότητα που είχαμε εάν ε, θέλαμε να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση η οποία θα ήταν όντω επικεντρωμένη στα συμφέροντα των, πολιτών, των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και χαίρομαι που σήμερα ψηφίσατε την έκθεση Γκρέσ. Συμπατριώτη μου είναι και πραγματικά έχει βάλει στον πυρήνα της έκθεσής του την πτυχή αυτή, την οποία υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά. Θα υπερασπιστώ λοιπόν αυτό το σημείο, στην ε, ομάδα των Επιτρόπων για την εσωτερική αγορά με τους οποίους θα συνεργάζομαι στενά. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι αυτή η ιδέα αναφέρεται στην έκθεση Γκρέσ που εγκρίνεται σήμερα το πρωί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέσ για την εξαιρετική του δουλειά και, να, και ελπίζω να επιτύχει μια, ένα εξίσου επιτυχές αποτέλεσμα και στην ε, ολομέλεια του επόμενου ε, μήνα. Επίσης συγχαρητήρια για την ε, υιοθέτηση της ε, έκθεσης HEAD η οποία θα δώσει μεγαλύτερο, ο, μεγαλύτερη όθηση στο scoreboard. Πρέπει να παρατηρούμε στενά πώς ε, υπηρετούν οι αγορές τους καταναλωτές και πώς μπορούν οι διάφορες δομές να, να αλλάξουν για να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Τώρα μελετώ το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το scoreboard. Ας πούμε Επεκτείνοντα και ενισχύοντα τι πληροφορίε που έχουμε ε, συλλέξει για το πώ δουλεύουν οι αγορές. Πέρα από αυτό, η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια σύσταση για τα, για τα παράπονα των καταναλωτών τον επόμενο μήνα που θα, δω, που θα δημιουργήσει τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούμε για να συμπληρώσουμε τα συγκρίσιμα δεδομένα που έχουμε από τους καταναλωτές. Κάθε χρόνο θα γίνονται δύο εις βάθους ε, μελέτες ε, για, την, για τους προβληματικούς τομείς και φέτος θα ολοκληρώσουμε τις μελέτες που γίνονται για την ε, αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και, το αγορά, και την αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Ε, ελπίζω να, να μου δώσετε την υποστήριξη που χρειάζεται ε, και σε οικονομικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ε, πολιτική μας και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή θα μας, θα μας βοηθήσει να, στοχο, να στοχεύσουμε καλύτερα τις αγορές και στην όλη οικονομική κατάσταση που αλλάζει αυτό περιλαμβάνει και τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα ψηφιακά προϊόντα, οι οικονομικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, να μην ξεχνάμε και τα οριζόντια θέματα της πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης κατανάλωσης θα συνεργαστώ στενά με την, με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ για τα θέματα τη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Την, ε, το τελευταίο, προηγούμενο μήνα, το, η, η Σύνοδο Κορυφή ε, για του ε, καταναλωτέ μα έφερε κοντά στο να δημιουργήσουμε να συνεργαστούμε με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και, και έκαναν, όπου έγιναν και πάρα πολλές συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, για την ενέργεια προσπαθούμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε προσκόμματα και στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτέ θα έχουν τη δυνατότητα και με τα, σωστά εργαλεία θα μπορούν να συγκρίνουν τι τιμέ και τι υπηρεσίε που λαμβάνουν. Θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τι ε, πρακτικέ που υπάρχουν και πώ μπορούμε να διαχειριστούμε τα παράπονα που, και πώ μπορούμε επίση να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά στον, στην απελευθέρωση του τομέα τη ενέργεια. Επίση, με τι σωστέ πληροφορίε που έχουμε, οι θα είναι πιο εύκολο να μπορούν να ε, συγκρίνουν και να περάσουν σε μια πιο βιώσιμη κατανάλωση ενέργεια. Τώρα, οι μεταφορέ. το, το χάος στι μεταφορές που δημιουργήθηκε από την, ε, από την ε, στάχτη πραγματικά έβαλε, στο, έβαλε, δοκίμασε του τους κανόνες για την εφαρμογή των κανόνων των, των δικαιωμάτων συγγνώμη, των καταναλωτών. Για το σχετικό πακέτο, εγώ θα συνεργαστώ με την Επίτροπο Ρέντι για να, εξασφαλίσουμε ότι ότι θα, υπάρχει καλύτερη, θα υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες για τους Ευρωπαίους επιβάτες. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει και φυσικά μεγάλη επίδραση και στο ε, περιβάλλον. Αλλά πρέπει να σα ε, διαβεβαιώσω ότι οποιαδήποτε δράση να λάβουμε στα πλαίσια τη βιώσιμη ανάπτυξη θα βασίζεται σε μια σαφή κατανόηση τη συμπεριφορά των καταναλωτών μα. Ε, τα ψηφιακά προϊόντα και οι υπηρεσίε στην αγορά επίση επηρεάζουν τη ζωή μα. Παρ' όλα αυτά, το ε, ρυθμιστικό πλαίσιο υπολείπεται κατά πολύ. Θα συνεργαστώ λοιπόν πολύ στενά με τον, με Αντιπρόεδρο Κρός για να ε, δημιουργήσουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, γίνεται όλο και περισσότερο, ε, η αγορά, η ηλεκτρονική αγορά γίνεται όλο και πιο ε, δεκτική, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και συμβάσεις online πιο φιλικές προς τους καταναλωτές και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ε, ιδιωτικότητα των καταναλωτών. Η οικονομική κρίση δείχνει πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει στην διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και μα δείχνει πόσο ε, άσχημη είναι η προστασία των καταναλωτών. Εγώ θέλω καταναλωτέ που να είναι καλύτερα προστατευμένοι στο μέλλον και, να, και που μπορούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη του στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών. Και γι' αυτό θα συνεργαστώ στενά με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Οι ε, μελέτε δείχνουν ότι οι καταναλωτέ επωφελούνται περισσότερο όταν είναι συγκεκριμένε οι πληροφορίε, εύληπτε και συγκρίσιμε. Θέλω να εξασφαλίσω ότι οι, δια, καταναλωτές θα λαμβάνουν τις απαραίτητε πληροφορίε και θα τις καταλαβαίνουν κιόλα. Πέρα από αυτό, θα φροντίσω να ε, προωθήσω ένα επίπεδο οικονομικής ε, ας εκπαίδευσης. Ε, το, το Dolcetta που είναι ένα εργαλείο online είναι μια πολύ καλή αρχή. Και επίσης μετά από την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου θα προετοιμαστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση σε υπηρεσίες επενδύσεων. Και η, επίσης η εφαρμογή ε, μέτρων έναντι των αθέμητων πρακτικών είναι κάτι που θα παρακολουθήσω. Ε, όπου και να ψωνίζει κανείς, είτε online είτε στα μαγαζιά, πρέπει να είναι ασφαλής. Αλλά σήμερα δυστυχώς έχουμε δύο παράλληλα προγράμματα επιτήρησης για τα, ουσ, ε, για τα, για τα αγαθά για τους καταναλωτές, ένα που το καλύπτει η Γενική ε, Οδηγία για την Ασφάλεια των ε, Προϊόντων και ένα για, με νέα που το καλύπτει η νέα προσέγγιση. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στους καταναλωτές και στις εθνικές αρχές και στους οικονομικούς ε, φορείς. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το, πρόγραμμα, το πρόβλημα, έχουμε αρχίσει να αναθεωρούμε την Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, προσπαθώντα να δημιουργήσουμε μια, ένα νέο ε, πλαίσιο για την ασφάλεια των προϊόντων. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε πιο σαφεί κανόνε, ε, πιο αποτελεσματική διαδικασία τυποποίηση και να αναλαμβάνουμε δράση πιο γρήγορα όταν υπάρχουν προβλήματα ή όταν βρίσκουμε επικίνδυνα, προγράμματα, επικίνδυνα προϊόντα συγγνώμη, στην αγορά. Και γι' αυτό θα Ήθελα και εσείς να κάνετε ακροάσεις ε, για την εποπτεία της αγοράς και την τυποποίηση. Ε, Βεβαίω, ε, οι αυστηροί κανόνε για την ασφάλεια των προϊόντων έχουν να κάνουν με την ε, στενή συνεργασία με του διεθνεί εταίρου μα, όπω η Κίνα και η ΕΠΑ. Και χαίρομαι που έχουμε αρχίσει να, ξε... να εξεργαζόμαστε τώρα, να διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων με τι Αμερικανικέ Αρχέ. Χτε έμαθα ότι μέχρι το τέλο του χρόνου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σε μια ανοιχτή οικονομία όπω η δική μα, θα πρέπει να επενδύσουμε όλο και περισσότερο στην συνεργασία με του εμπορικού μα εταίρου. Ε, στο μελλοντικό μου ταξίδι στην Κίνα ε, θα, γίνει, θα έχω αυτό το στόχο στο μυαλό μου για να του πείσω για το πόσο μεγάλε είναι οι απαιτήσει των Ευρωπαίων καταναλωτών για ασφάλεια. Είναι σαφέ ότι οποιαδήποτε νομοθεσία δεν είναι αχρηστή εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Η κοινοποίηση του, της Κομισιόν του προηγούμενου Ιουλίου καταδεικνύει τους τρόπους με τον οποίο μπορεί η, εφαρμογή να γίνει πιο επιτελεσματική και συνεπής με, στα, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτέλους τώρα η θεωρία πρέπει να γίνει πράξη. Αυτό βέβαια απαιτεί και πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς για να μπορέσει να γίνει η κατάλληλη δουλειά από αυτούς που θα την κάνουν. Κατανοώ ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Επιτροπή HED, για την η Χέντι, η Επιτροπή σα έκανε, ε, μελέτησε την ιδέα να κάνει μία ακρόαση με, ε, τους, με νομοθέτες, με ε, όσου ασχολούνται με το θέμα αυτό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πραγματικά θα ήταν ένα, μια μοναδική ευκαιρία για, την, για μια συζήτηση που χρειάζεται να γίνει για την εφαρμογή και που θα εξασφαλίσει ότι αυτό σε αυτό το θέμα θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα. Τι κάνει όμως ο καταναλωτή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ θέλω να, οι καταναλωτέ να έχουν την εμπιστοσύνη και τα εργαλεία για να δράσουν. Θα ε, απαντήσω στο αίτημά σα και θα παρακολουθήσω την ε, πράσινη βίβλο για την ε, αναθεώρηση για τους καταναλωτέ. Έχουμε ήδη ξεκινά, ξεκινήσει με τον Επίτροπο Αλμούνια και την κυρία Ρέντινγκ τη δημιουργία ενό ε, ε, ε, αποτελεσματικού πλαισίου για το θέμα αυτό και η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση τον, το φθινόπωρο. Ε, πιστεύω ότι τέτοιε διαβουλεύσει είναι ωφέλιμε για του καταναλωτέ και θα με διευκολύνει και εμά να προχωρήσουμε γρήγορα προ τα μπρο με τι διάφορε προτάσει που έχουμε. Επίσης ε, η διαβούλευση αυτή είναι μια ευκαιρία για να ε, αφήσουμε τις, ε, τους δισταγμούς και που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση των δικών μας τύπων ανέτη των Αμερικανικών. Και επίσης είναι πολύ νωρίς ακόμη να μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικέ νομοθετικές προτάσεις. Αλλά εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα αφοσιωθώ στο θέμα αυτό και σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο θα έχουμε μια πρόταση την οποία θα σας υποβάλουμε για να τη μελετήσετε. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι η δουλειά αυτή μπορεί να ξεκινήσει με, την, με το ψήφισμα για την, με το Alternative Dispute Resolution, το οποίο είναι ένας τομέας κλειδί για οποιοδήποτε σύστημα ε, αποκατάστασης θέλουμε, ζημιών που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ε, μπορεί να δημιουργήσει ένα φτηνό, απλό και άμεσο τρόπο να αποκατάσταση των ζημιών έναντι των καταναλωτών και να ε, ε, λύσει προβλήματα μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων. Κλείνοντα, ε, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να σα αναφέρω πώ ακριβώ θα συνεργαστώ με του συναδέλφου επιτρόπου και πώ μπορώ να πώς θα προχωρήσω στο δικό μου τομέα για να έχουμε απτά και φιλόδοξα αποτελέσματα για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Θα έρθω και πάλι στην Επιτροπή σα πριν το τέλο του έτου, όσο θα εξελίσσεται η δουλειά μα, με μια, μια, καταγραφή των δράσεων που θα περιλαμβάνουν όλα τα ωφέλη που θέλει να επιτύχει η Κομισιόν για την προστασία των καταναλωτών στα επόμενα πέντε χρόνια. Επίση, σύμφωνα και με τις, εκθέσει τη κυρία εκθέσεις της κυρίας Χέντ, του κυρίου Γκρέσ και του κυρίου Αρία. η στρατηγική αυτή θα δείξει ότι κατά την άποψη της Κομισιόν οι καταναλωτέ μπαίνουν στον πυρήνα τη της αγορά αγοράς και η δική τους ευημερία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εσωτερική αγοράς. Βεβαίω, θα... Ε, θέλω να ακούσω και τις δικές σας ε, ιδέες ε, σε σχέση με αυτά που είπα σήμερα και βεβαίω. Ε, βασίζουμε στην ε, συνεργασία και την υποστήριξή σας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε όντως να φέρουμε ωφέλη για τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ. Uh, well, thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ περιεκτική και φιλόδοξη η παρουσίασή σας, όπως και το πρόγραμμά σας και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας. Αναφερθήκατε σε πολύ, σημαντικά, σε πολύ σημαντικές εκθέσεις ε, δικές μας, ε, της κυρία, την έκθεση HED, Greg. Ε, Θα κάνω τώρα την εξής πρόταση, συνάδελφοι, για το χρόνο μιλίας. Θα ήθελα να προτιμήσουμε εκείνους που δεν μίλησαν προηγουμένως. Εννέα μιλητές, μισή ώρα. 1,5 λεπτό έκαστος. Και η κυρία Ρούλε επίσης θέλει να πάρει το λόγο, οπότε 10 είναι οι ομιλητές μας συνολικά. Πέντε ομιλητές τη φορά και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος. Έχω και τον κύριο Ντε Η κυρία Κοράτσα. Πήρε το λόγο, νομίζω πρώτη απέσπασε την προσοχή μου. Ροσφόρ, Ταραμπέλα. Και μετά θα δούμε, θα αποφασίζω για τη σειρά των υπολείπων ομιλητών. 1,5 λεπτό όμως. Πρώτα η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και μετά ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σαφές σας όραμα. Γιατί η ευημερία των πολιτών και οι καταναλωτές είναι στο, είναι στο επίκεντρο της προσοχής σας. Είπατε ότι γυρίσατε μόλις από τι Ηνωμένε Πολιτείε και είπατε ότι δεν ε, ε, θα αρθεί απαγόρευση των ε, κοτόπουλων που έχουν καθαριστεί με χλώριο. Νομίζω ότι εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο... Συγγνώμη που σας, διακόπτει, σας διακόπτει λέει ο, πρό, πρόεδρος. Μιλάμε για το πρόγραμμα εργασίας της συγκεκριμένης της συγκεκριμένης ε, ε, επιτροπής. Αυτά που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά δεν είναι το αντικείμενό μας αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να ρωτήσουμε τον κύριο Ντάλι για τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Μα συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι βασική η δουλειά μα ε, η προστασία του καταναλωτή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να απαντήσει στο ερώτημά μου. Ναι, είναι, αλλά είναι και επίκεντρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, τη δουλειά Επιτροπή Περιβάλλοντο. Οπότε, αν θέλει ο κύριο Ντάλι να απαντήσει, καλώ. Αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω τι σχέση έχει. Να συνεχίσουμε. Η κυρία Βανιού. Κυρία Βερνιό. Faire attention aux questions que je pose parce que je voudrais pas trop θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να μην πλατιάσω. Μιλήσατε πολύ για την πολιτική των καταναλωτών και πιστεύω ότι μπορούμε να αναβιώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη πολιτική αυτή. Μιλήσατε για την, για την ετικετοθεσία ε, στα τρόφιμα. Εγώ προσωπικά ήμουν εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Έχουμε ακόμη πολλέ φαιέ ζώνε αόριστε στο τομέα αυτό, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη ετικετοθεσία δεν θα λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχει εκστρατεία ενημερωτική από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ε, επικράτεια. Έχουμε παρκή οικονομικά μέσα για να το κάνουμε αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για έλλειψη διαφάνεια στι ε, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Πάρα πολύ επίκαιρο αυτό που είπατε. Σήμερα το πρωί το ανέφερε και ο κύριο Μπαρνιέ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επιγόντω πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μία ακόμη ερώτηση ενδεχομένω να μην είναι τόσο σχετική, ε, κύριε Πρόεδρε, αλλά ήμουν συντάκτρια γνωμοδότησης ε, για, τις διασυνοριακές, ε, για τη διασυνοριακή ιατρική φροντίδα και η Ισπανική Προεδρία ήθελε να ε, ξανασυζητηθεί το θέμα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτό το, αυτά τα θέματα ε, βεβαίως, ε, γιατί έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Ε, η ασφάλεια των τροφίμων και τα κατόπουλα δεν, μας, ε, δεν είναι στο επίκεντρο βέβαια της δουλειάς μας, γι' αυτό ήμουνα με την κυρία Βερνιό τόσο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας είπατε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την δική μας Επιτροπή. Ε, συμφωνώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, την προσπάθειά μας όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα ε, να νομίζουν ότι είμαστε απλώς επιθετικοί μαζί τους με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Κρίμα όμως που το κείμενο που αφορά το δικό σας χαρτοφυλάκιο και το πρόγραμμα εργασίας για το 2010 είναι προϋπόθεση, έχετε θέσει ως προϋπόθεση γι' αυτό είναι διαβούλευση. Έχω λίγο την εντύπωση ότι τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Μιλήσαμε για μια συλλογική ε, προσέγγιση, η οποία είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάποια πράγματα που είπατε. Έχουμε τις συνέπειε τη ηφαιστιακή έκρηξη, τεράστια κρίση που έπληξε τους καταναλωτές και καταλαβαίνω ότι ο κύριο Κάλλα ενδεχομένω να πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό του συντονισμού των μεταφορών, αλλά μιλάτε πολύ συχνά για την προστασία των καταναλωτών. Και τώρα έχουμε μπροστά μας μία ακόμη κρίση, δεν ξέρω, μπορεί σε μερικές εβδομάδες το απέφχομαι, αλλά μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι ένα τέτοιο θέμα, ένα τεράστιο νέφος που θα ε, μπλοκάρει εντελώς τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Τι θα κάνουμε ώστε Δεκάδε χιλιάδε Ευρωπαίοι να μην βρίσκονται, να μην έχουν ξεμείνει σε διάφορα αεροδρόμια. Μήπω θα έπρεπε να έχουμε κάποιο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκό, να δούμε ε, πώ μπορούμε να τους βοηθήσουμε, βέβαια σεβόμενοι την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει κάπως να τους βοηθήσουμε, να δώσουμε μία όθηση. Αυτό είναι κάτι το απαραίτητο, αν λέμε τώρα, και το απέφχομαι επαναλαμβάνω, ε, υπάρξει μία τέτοιου είδους κρίση ξανά. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι, όπως είπε και ο κύριος Ροσφόρ, ε, Πάρα πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν ε, στους ε, πολίτες λόγω της ηφαιστειακής έκρηξης. Πρώτο πρόβλημα, πλήρη έλλειψη συντονισμού μεταξύ αρμοδίων αρχών ε, της, μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόβλημα για τις αεροπορικές εταιρείε. Τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε επίση και τον κανονισμό 2061 του 2004 που αφορά την ακύρωση των πτήσεων και τη σχετική αποζημίωση των ε, ε, ε, των επιβατών, μήπως θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε αυτήν την οδηγία η οποία είναι 20 ετών και να την τοποθετήσουμε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασία δεδομένων των προβλημάτων που ήδη υπήρξαν και που μπορεί να υπάρξουν ξανά και στο μέλλον. Δεύτερον, το είπατε και εσεί. το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας ε, όσον αφορά τις συνέπειε τη απελευθέρωση που τους γνωρίζουμε και στην ενέργεια και στις ταχυδρομικέ υπηρεσίε, Θα υπερασπιστείτε την ιδέα μια αξιολόγησης ε, του αντικτύπου της απελευθέρωσης για τον ίδιο τον καταναλωτή. Μα είναι σαφές ότι όλες αυτές, ε, όλη αυτή η απελευθέρωση έγινε, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη σε σχέση με τις συνέπειες αυτής της απελευθέρωσης. Είναι γεγονός ότι πλέον ε, είναι πιο ακριβές ε, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, λιγότεροι εργαζόμενοι. Ελπίζω οι καταναλωτές βέβαια να εξυπηρετούνται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει έχετε σκοπό να ε, υπερασπιστείτε μια τέτοιου είδου αξιολόγηση στον πρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στήλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ Επίτροπε ε, Ντάλι ε, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Μιλήσατε για, τον, ε, για, για την χρηματοπιστωτική κρίση, για τους σχετικούς κανονισμούς. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μπαρνιέ το έθεσε επίσης και το συνέδεσε και με το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Πώς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μπαρνιέ για το θέμα αυτό, γιατί είναι ζωτική σημασία. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι σημαντικές για τους πολίτες ε, σε καθημερινή βάση. Επίσης, ε, μιλήσαμε για τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν ξέρω αν είχατε συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά είναι και αυτό κάτι το πολύ σημαντικό. Μήπως θα, έπρεπε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Ροσφόρ μίλησε για τα δικαιώματα των επιβατών. Θέλουμε να έχουμε και τη νέα οδηγία για τους ε, ε, ταξιδιώτες. Κάποιες εταιρείες τα κατάφεραν καλά, Κάποιε εταιρείε δεν τα κατάφεραν καλά και λαμβάνουν επιστολέ αυτή τη στιγμή σε σχέση με την αποζημίωση των επιβατών εννοώ και με τη συμπεριφορά προ του επιβάτε. Πώ θα εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε μα δεν θα έχουν τέτοιου είδου προβλήματα ε, με μια αεροπορική εταιρεία που θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο, περισσότερα για έναν άνθρωπο που έχει ξεμείνει σε ένα αεροδρόμιο και σε άλλε περιπτώσει, ούτε νερό δεν του έδωσαν στους ανθρώπου. Πώς θα γίνει λοιπόν Όλο ο κόσμο, πολλοί άνθρωποι περιμένουν μια ολόκληρη χρονιά για να ε, πάνε διακοπέ με ένα πακέτο που έχουν κλείσει καιρό και έχουν αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσουν. Και κάτι ακόμη. Έχω διαβάσει μερικά πράγματα για τα δικαιώματα των Τζον στον Αμερικανικό τύπο κλπ. Νομίζω ότι είναι σημαντική η συνεργασία μας με τους Αμερικανούς. Ε, υπάρχει και μία πρόταση συνεργασία σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Εξαιρετική ιδέα και θα ήθελα να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που συζητήσατε το εν λόγω θέμα. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου πείτε λίγο περισσότερα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ντάλι να απαντήσει στο πρώτο πακέτο ερωτήσεων μεγάλη ποικιλία θεμάτων, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε να απαντήσετε σε όλα. Να ξεκινήσουμε με τα χλωριωμένα κοτόπουλα. Αυτό που συζητούσαμε και εδώ και καιρό με τη ΣΥΠΑ ήταν οι επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον, τις αντιμικροβιακές το αντιμικροβιακού αυτού πλησίματος των, των πουλερικών. Εμείς έχουμε κάποια πρότυπα βάσει των οποίων μεγαλώνουν τα δικά μας ζώα και βεβαίως και υπάρχουν αντίστοιχα πρότυπα. Εμείς επιμένουμε ότι θέλουμε να έχουμε τα καλύτερα πρότυπα σε όλη την αλυσίδα της διατήρησης ζώων και σε ό,τι μας αφορά αυτό μας δίνει ένα ασφαλές προϊόν στο τέλος και ένα ποιοτικό προϊόν. Ένα δηλαδή προϊόν που είναι πολύ καλύτερο αν δεν είχαμε ακολουθήσει αυτά τα πρότυπα. Από το αν δεν είχαμε ακολουθήσει αυτά τα πρότυπα. Τα είδη δεν λαμβάνονται τόσο πολύ υπόψη. Έχουμε τα σφάγια, έχουμε τα πουλερικά τα οποία την χάνουν καθαρισμού με αυτά τα αντιμικροβιακά προϊόντα για να είναι ασφαλή για κατανάλωση. Πολλοί καταναλωτές έχουν ε, παραπονεθεί γι' αυτό και πολλές χώρες έχουν σταματήσει και τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων στην Ευρώπη. Εμείς κάναμε τη δική μας αξιολόγηση της κατάστασης. Ακόμη θέτουμε πολλά ερωτήματα στους Αμερικανούς ομολόγους μας. Έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα με τους Αμερικανούς, το οποίο θα τηρήσουμε. Και η φάση στην οποία βρισκόμαστε είναι η εξή. Έχουμε στείλει μια επιστολή, ένα κατάλογο μάλλον, ένα ερωτηματολόγιο, στους ε, Αμερικανούς κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να αμβλύνουν και να εμπλουτίσουν το επιστημονικό φάκελο, τον επιστημονικό φάκελο που του έχουμε αποστείλει. Στι συζητήσει που έκανα χτε και προχτέ, οι Αμερικανοί δεν είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Αλλά εξηγήσαμε ότι αυτό εμεί το χρειαζόμαστε. Είναι σημαντικό για μα. Και αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε. Για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, φυσικά οι Αμερικανοί καλωσορίζουν το γεγονό ότι όλη αυτή η ιδέα ότι η Ευρώπη μπλόκαρε τον εαυτό της ουσιαστικά με τους μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς τώρα τελειώνει. Εγώ κατέστησα απόλυτα σαφές ότι κατά δική μας άποψη είμαστε υπέρ της κοινοτομίας, εγώ είμαι υπέρ της κοινοτομίας, αλλά υπεύθυνη κοινοτομίας. Η υπεύθυνη κοινοτομία για μένα, και χαίρομαι που το συζητούμε σήμερα, η υπεύθυνη κοινοτομία λοιπόν σημαίνει ότι εγώ θέλω να εξασφαλίσω ότι η, η κοινοτομία και τα προϊόντα που ε, παράγονται βάσει αυτής μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες. Και σε αυτό θα επιμείνω, σε αυτή τη συζήτηση για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Και επίσης, ζήτησα από τους Αμερικανούς και θα συμφωνήσουν ε, να κάνουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων, των αποτελεσμάτων που έχουν εδώ και μια δεκαετία. Αυτοί έχουν εδώ και μια δεκαετία εμπειρία στην, ε, στο θέμα αυτό. Οπότε θέλουμε πληροφορίες εμείς από αυτούς και αξιολογήσεις, εκτιμήσεις για παρατηρήσεις που έχουν κάνει από ανεξάρτητους φορείς, όχι από τις ε, μπλεκόμενες εταιρείε δηλαδή, για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που είχαν, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ε, απενοχοποιήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση και να μπούμε στην ουσία. Οι Αμερικανοί ε, μας είπαν ότι θα, συμφω... θα μας δώσουν τις πληροφορίες και είναι σε επαφή με τη ΣΑΝΚΟ για να αρχίσουν να μας στέλνουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή είναι η τάση και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Ε, επισήμανση τροφίμων. Σημαντικό. Αν εγώ θέλω να δω τι θα ήθελα να έχω επιτύχει στο, στο τομέα των καταναλωτών, η απάντηση θα ήταν θα ήθελα να έχω ε, ενισχύσει τον ε, καταναλωτή, έτσι, να τον έχω βοηθήσει έτσι ώστε οι αποφάσεις του και οι ανάγκες του να επηρεάζουν την πολιτική μας. Αυτό είναι ο δικός μας στόχος. επ' αυτού εργαζόμαστε εμείς για τους καταναλωτές. Οι πληροφορίες, εντάξει, είναι σημείο κλειδί. Γιατί για να υπάρξει μια ε, σωστή απόφαση πρέπει κανείς να έχει την, απόλυτη, την πλήρη ενημέρωση. Οπότε εμείς θέλουμε να δώσουμε στους καταναλωτές όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Εγώ οικονομολόγος είμαι στο επάγγελμα, και ξέρω ότι τα πάντα έχουν ένα κόστος. Όλα έχουν μια τιμή. Οπότε πρέπει να είναι πολύ ισόρροπα τα πράγματα. Πρέπει να είναι πολύ ισόρροπες οι ε, προτάσεις μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να αρχίσουμε να δίνουμε έτσι, πληροφορίες αβασάνιστα ε, στους καταναλωτές. Ε, πρέπει να είναι κατανοητά αυτά που τους λέμε. Πρέπει να ξέρουν πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι κάνοντας τις, για τους εαυτού τους πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι κάνοντας τις ε, επιλογές τους. Θέλουμε λοιπόν έτσι μια συνολική προσέγγιση και με τις υπηρεσίες μας ξεκινούμε τη διαδικασία τώρα για να αναλύσουμε το κόστος και τα ωφέλη όλων αυτών των τομέων. Συγγνώμη αν μακρηγορώ, αλλά ε, σε μία από τι συναντήσει με, την, με τη ΣΥΠΑ ε, ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο για την ε, ε, έξυπνη νομοθεσία, έξυπνη ρύθμιση ε, που έχουν να κάνουν και με, με την οικονομική πτυχή και οι οποίοι έχουν συμπεριλάβει την αξιολόγηση επιπτώσεων και έχουν δώσει μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση επιπτώσεων. Δηλαδή δεν αξιολογούν απλώς το κόστος και το οικονομικό όφελος, αλλά βάζουν και τον ε, παράγοντα άνθρωπο στην όλη εξίσωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Σάνκο ήδη ε, το έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αυτό, δεν είναι δηλαδή καινούριο. Ε, οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν έχει νόημα να βάζουμε πληροφορίες στις συσκευασίες που δεν μπορούν να τις καταλάβουν οι καταναλωτές η ε, εκπαίδευση σε εισαγωγικά των καταναλωτών είναι καλή. Είναι το, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Βλέπετε τώρα στις, στα μπουκάλια, ας πούμε, ε, του, των νερών, τι λέει. Λέει πόσα μέταλλα έχει, πόσα γνωστοιχεία. Ναι, αλλά αυτά τα μέταλλα εμένα τι μου κάνουν στη δική μου την υγεία. Mm. Αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά που διαβάζουμε. Γιατί αλλιώ τι νόημα έχει. Έχουμε κάνει κάποια ενημερωτικά προγράμματα με 15 κράτη-μέλη και θα ξεκινήσουμε και με τη Ρουμανία τον επόμενο χρόνο, άλλο ένα τέτοιο πρόγραμμα, αρκετά δαπανηρό πρέπει να πω. Και εδώ θα πιέσουμε ώστε να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων που είναι τόσο σημαντικά για να επιτύχουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί να επιτύχουμε. Και επίσης ε, να σας πω και κάτι άλλο. Ε, επιμένω στις δικές μου υπηρεσίες ότι η διαδικασία ε, προπολογισμού η δική μας δεν θα είναι η συνήθις γραφειοκρατική δημοσιοϊπαλληλική διαδικασία. Όχι πόσα πήραμε πέρσι, πόσα θα ζητήσουμε του χρόνου. Να, υπάρχει, να είναι στοχοθετημένη ανάλογα με το πρόγραμμα. Δηλαδή θα ποσοτικοποιήσουμε πόσο θα κοστίσουν τα προγράμματα, θα ποσοτικοποιήσουμε όλα τα προγράμματα τα οποία ξεκινάμε και τα οποία μας έχει ζητηθεί να ξεκινήσουμε, θα τα, θα τα κοστολογήσουμε και μετά θα υπάρξει η πολιτική απόφαση για το ποια είναι τα προγράμματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με, το, με τη γραμμή που θα θέσουμε ως όριο. Διασυνοριακή υγεία. Το είπα ότι θα συνεργαστώ με την Ισπανική Προεδρία για τη διασυνοριακή υγεία. Το κάνω ήδη. Και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι έχει υπάρξει αρκετά καλή κινητικότητα, αρκετή κινητικότητα από την Ισπανική Προεδρία για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Στην τελευταία άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας στην ε, Μαδρίτη ε, την τον Υπουργό στην Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ισπανική Προεδρία ε, μας παρουσίασε ποια είναι, ποιο είναι το σκεπτικό τη για το πώ μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Και παρόλο που λάβαμε αρκετά θετικά σχόλια από πολλά κράτη-μέλη, και τα υπόλοιπα μέλη που αποτέλεσαν την, ε, τη μειοψηφία η οποία μπλόκαρε το θέμα, κινήθηκαν και αυτά. Ακόμη δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική απόφαση βέβαια, γιατί πολλές χώρες, και κατανοητό είναι, ε, ήταν αρκετά συντηρητικέ, μα είπαν ότι έχουν επιφύλαξη, πρέπει να το, να το μελετήσουν, πρέπει να πάνε στου εμπειρογνώμονε. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι αρκετά φιλόδοξη, είναι αρκετά θετική. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει όντω να μετακινηθούμε και εμεί προ αυτή την κατεύθυνση. Συλλογική αποζημίωση. Αποκατάσταση. Ε, η συλλογική αποκατάσταση είναι όντως ε, προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Συλλογικά κινούμεθα. Καταρχήν για να κατανοήσουμε σε βάθος όλα τα σημεία και με τον Αλμούνια και με τη Ρέντινγκ γιατί δεν θέλουμε εντάξει θα υπάρξουν δύο ε, νομοθετικά κείμενα το ένα με βάση τους καταναλωτές και το άλλο με βάση το εμπόριο και τα δύο θα αφορούν την συλλογική αποκατάσταση των ζημιών, αλλά να μην υπάρχουν και αμφισημίες μεταξύ των δύο, έτσι, ή να μην ε, πατάει το ένα στα χωράφια του άλλου. Οπότε θα γίνει η διαβούλευση αυτή και ελπίζω μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους να μπορέσουμε να σας υποβάλουμε νομοθετική πρόταση. Τώρα, το ηφαιστειακό σύννεφο. Καταστροφή όχι μόνο γιατί πολλοί από εμά και ο υποφαινόμενος δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη δουλειά τους με αρκετές συνέπειες που θα τις δούμε αλλά και λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Οι πολίτες πραγματικά υπέφεραν υπέρμετρα με αυτό το γεγονός. Η Κομισιόν κινήθηκε γρήγορα και προσπάθησε να δει ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθορίζοντας ποια είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Βέβαια, εντάξει, κάποιοι μεταφορείς προσπαθούσαν να το παίξουν ε, δύσκολοι, αλλά τα δικαιώματα των πολιτών είναι αυτά που είναι, τα δικαιώματα των καταναλωτών έχουν, οι καταναλωτέ έχουν δικαίωμα στην αποζημίωση, ε, δικαίωμα σε ε, στέγαση ανάλογα με τις ημέρες του, που κράτησε το φαινόμενο, ενημέρωση και εμείς επιμείναμε σε όλα αυτά. Και τα κέντρα, οι ενώσεις των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη μας δίνουν τώρα ε, feedback για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αντιμετώπισαν. Βεβαίως εμείς καλωσορίζουμε πάντα οποιαδήποτε συμβολή από οποιονδήποτε που έχει υποφέρει λόγω αυτή, αυτής της κατάστασης, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ο αριθμό των παραπώνων οχταπλασιάστηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κινούνται τα πράγματα. Την Τη Δευτέρα η Κομισιόν ε, ε, ε, οργάνωσε μια διάσκεψη για του νομοθέτε, ώστε να συζητήσει επιχειρησιακά θέματα και ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα ήταν τι κάνουν οι επιβάτε όταν δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τι αεροπορικέ εταιρείε για να κανονίσουν τα ταξίδια του από μόνοι του. Οι αεροπορικέ εταιρείε παραβιάζουν τον νόμο σε τέτοια περίπτωση γιατί οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα στην αποζημίωση του κόστους που έχουν ήδη πληρώσει. Πρέπει να πω ότι η Κομισιόν προσπαθεί να ενισχύσει τις αεροπορικές εταιρείες για, τα, για τις απώλειές τους, αλλά ε, βάζουμε προποθέσεις. Οποιαδήποτε βοήθεια δοθεί βασίζεται και στο κατά πόσο συμμορφώθηκε και σεβάστηκε την νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών η εταιρεία αυτή. Αν δούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν, δεν συμμορφώθηκε με την, με την νομοθεσία, δεν δικαιούται οποιαδήποτε είδους, οποιαδήποτε είδους βοήθεια. Για την ενέργεια, ναι, έχουμε επικεντρωθεί στην ενέργεια φέτος και όπως είπα στην ομιλία μου, ένα από τα θέματα, ένα από τα scoreboards που θα βγει φέτος είναι για την, ε, λιανική, για την αγορά λιανικής ε, στην ενέργεια. Γιατί λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί αν δεν λειτουργεί και όταν θα έχουμε τις πληροφορίες αυτές, θα τις συζητήσουμε και θα αναλάβουμε δράση αναλόγως για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι υπολειτουργούν στον τομέα αυτό. Για τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό. Καταστροφή τα τελευταία δύο χρόνια σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, η οικονομική ύφεση που περνάμε οι οικονομικέ ε, υπηρεσίε είναι διπλές. Υπάρχουν αυτοί που δανείζονται και αυτοί που επενδύουν. Και για του δύο πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, μεταρρύθμιση για το πώς, μπορούμε να διαχειριστούμε τους καταναλωτές για τους δύο αυτούς τομείς. Υπάρχει ανάγκη για πληροφόρηση που να είναι σαφής, που να είναι ξεκάθαρη, που να είναι συγκεκριμένη και η δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τα δεδομένα μεταξύ του ενός χρηματοπιστωτικού και του άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Θα θέλαμε λοιπόν να δοθεί περισσότερη έμφαση, ειδικά σε ό,τι αφορά το δανεισμό και μεγαλύτερη ευθύνη από, τον, από τους δανειστές. Να εξασφαλίσουμε ότι ο δανειζόμενος μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο που λαμβάνει. Αυτή η πίεση πρέπει να ασκηθεί έτσι ώστε να δημιουργηθεί ε, μια πιο φιλική προς το χρήστη προσέγγιση για, από τους δανειστές. Πριν πάω στις ε, είπα, έκανα μια, έδωσα μια συνέντευξη και με ρώτησαν βεβαίω και για τα δικαιώματα των ζώων και μου είπαν και για αυτά τα, το πλήσιμο με τη χλωρίνη κτλ. Ε, είναι θέμα δοκιμό, για το θέμα δοκιμών ε, σε ζώα για τα καλλιντικά. Εγώ είπα ότι αυτή τη στιγμή, τη χρονική, δεν θέλω να επεκτείνουμε τις, απο, τις παρεκκλήσεις ως προς αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε να, υπάρξει κάποιο να υπάρξουν αντικατα... υποκατάστατα. Νομίζω ότι έχω καλύψει τις ερωτήσεις σας. Λυπάμαι που μακρηγόρησα. Uh, uh, uh, μας είπατε και ορισμένα πράγματα που ήταν ε, εκτός της σημερινής μας, ε, του σημερινού μας αντικειμένου της συζήτησης, αλλά η κυρία Κοράτσα έχει φύγει. Εν πάση περιπτώσει απαντήσατε στο ερώτημά σας, της. Ο κύριος Αράγιος που είναι πρώτος ε, στην στον κατάργο των ομιλητών. Θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκρέκ είναι μετά. Και μετά έλεγα να περάσουμε στους συντονιστές με αντίστροφη σειρά από αυτήν που ακολουθούμε συνήθως. De Jong, Ρούλε, Μπουζόι, Κέπχαρτ και Σφάμπ. Μπορεί να μην θέλετε να πάρετε όλοι το λόγο γιατί μπορεί να σας κάλυψε με τις απαντήσεις του ήδη ο Επίτροπος αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι τις 6 παρατέταρτο γιατί μετά έχουμε και μία έκθεση να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο Ντάλι γιατί μας αφιέρωσε μέρος του χρόνου του. Μιλήσαμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο και βλέπω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι βασικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του. Εργαζόμαστε για μία έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία πλούστευσης και εναρμόνισης έτσι ώστε να άρουμε τα προσκόμματα μέσα στα πλαίσια μιας ψηφιακής ενίας αγοράς έτσι ώστε να προωθήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην καθημερινή μας ζωή σαν κάτι το απόλυτα οικείο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκρέχ. Ευχαριστώ πολύ. Όλα όσα αναφέρατε στο πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, καταναλωτών και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να επιτύχετε τους στόχους ε, αυτούς. Όμως, έχω ένα πρόβλημα. Αν όλες αυτές οι προτεραιότητες για τους καταναλωτές και η διαχείριση όλων αυτών, γιατί μιλήσατε για διάφορες πρωτοβουλίες, ε, είπατε ότι κάποιες είναι προσωπικές δικέ δικές σας, ε, άλλες προέρχονται από άλλες γενικές διευθύνσεις, από άλλους επιτρόπους. Συμφωνώ όντως ότι έχουμε πολλές προτεραιότητες, αλλά ανησυχώ μήπως στο τέλος δεν επιτύχουμε τίποτε από όλα αυτά. Υπάρχει μια κοινή στρατηγική την οποία να έχετε προγραμματίσει και τις οποίες εσείς θα είστε ο συντονιστής, όπως ζητήσαμε εμείς, ώστε τελικά να μην υπάρχει κάτι το κατακαιρματισμένο μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και χωρί καμία αξία για τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος De Jong. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Συμφωνώ με τον κύριο Ταραμπέλα που έθεσε το ερώτημα σχετικά με την απελευθέρωση των ε, ταχυδρομείων θέσαμε και προφορική ερώτηση για τον αντίκτυπο του ζητήματος αυτού και στους εργαζομένους και στους πολίτες. Υπάρχει άλλωστε και μία αναστολή της και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Έχουμε ακούσει πολλά παράπονα από τις επιχειρήσεις ε, Πολλέ φορέ ε, σα έρχεται ένα email, σα ζητούν να δώσετε τα στοιχεία σα και τελικά έχετε υπογράψει μια σύμβαση χωρί καλά-καλά να το καταλάβετε. Αυτό είναι παράνομο όπω καταλαβαίνετε. Ποιο μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί όλο και επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση τον τελευταίο καιρό. επίση η σημασία των ε, ε, οργανισμών καταναλωτών, των ενώσεων καταναλωτών, που έχουν εξαιρετικέ ιδέε, αλλά παραπονιούνται συνεχώς και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους ότι η επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εύκολη. Μήπως θα μπορέσετε κάτι να κάνετε ώστε να μπορούν πιο εύκολα να έρχονται σε επαφή μαζί σας οι καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Jong. Πρέπει να πω, για να με δίκαιος με την κυρία Κοράτσα Μπίλς, ότι Ούτε η απελευθέρωση των ταχυδρομείων έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητούμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουμε γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή ε, ε Μεταφορών. Η κυρία Ρούλε. Εντυπωσιάστηκα κύριε Νταλή από, την, ε, από το εύρος και την ταχύτητα με την οποία εργάζεστε. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Για τα θέματα των, ε, των ε, γενετικώς μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, αλλά το πώς έχετε βάλει στον πυρήνα τη συζήτηση και των ε, πράξεών σας τους καταναλωτέ είναι εντυπωσιακό. Για τη νέα προσέγγιση και την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων, πραγματικά υπάρχει μεγάλη σύγχυση στα κρατημέλη για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σας, να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ, εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Η προσέγγιση σας από την αρχή είναι καλή. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε χώρες όπως η Κίνα και η ε, ΕΠΑ να, να τις ε, κάνουμε να συμμετάσχουν γιατί στο τέλος συνήθως ε, εμείς σκεφτόμαστε πολύ αργά να δούμε ποια είναι τα δικά τους προβλήματα και ποια είναι τα δικά τους πρότυπα αλλά αν γίνει αναθεώρηση ίσως μεταρρύθμιση, ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να δούμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες και αν αυτό λειτουργεί να το υιοθετήσουμε κι εμείς. Επίσης ε, ζήτησα τον ε, λόγο για τον προπολογισμό, γιατί είπατε ότι θέλετε να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και αυτό είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή φέτος Ατυχώ είμαι η εισηγήτρια για την Επιτροπή μα για τον προπολογισμό και πάντα η εμπειρία μου είναι ότι το τομέα των καταναλωτών διαγράφεται πάντα από το Συμβούλιο. Οπότε η προσφορά μου προ εσά για συνεργασία ισχύει έτσι ώστε για να έχουμε και για τον τομέα αυτών των καταναλωτών του πόρου που χρειάζονται. Για πιλωτικά προγράμματα α πούμε, τα οποία ούτω ή άλλω είναι λογικά και σκόπιμα να υπάρχουν και τα έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή αυτή και για το Φόρουμ για την Ιστορική Αγορά ε, και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, εδώ πρέπει να γίνουν ε, δημόσιες ακροάσεις και για την ε, συλλογική αποκατάσταση ζημιών, που επίσης είναι καλό, και για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που επίσης είναι καλό. Και αν έχετε και άλλες προτάσεις, θα σας ήμουν ευγνώμων γιατί και εμεί μπορούμε να κινητοποιηθούμε σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει που κάνουμε για τον προπολογισμό. Και κάτι άλλο για, τις για την πληροφόρηση. Συμφωνώ απολύτω 100% μαζί σα Είναι καλό εάν η Κομισιόν κάνει κάποια στιγμή μια πρόταση, γιατί από τη μία έχουμε την εικόνα των ενημερωμένων πολιτών και από την άλλη καταναλωτών και από την άλλη ξέρουμε ότι οι καταναλωτέ ε, πραγματικά ε, τους πλημμυρίζουν οι πληροφορίε. Πρέπει να είναι και λίγο ε, οι πληροφορίε που λαμβάνουν. Υπάρχει και η σχετική οδηγία και το θέμα αυτό προκύπτει πάντα. Και όταν η Κομισιόν, θα, αν η Κομισιόν ήθελε να αφουσιωθεί στο θέμα αυτό, καλό θα ήταν να έχουμε α πούμε, κάποιε κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς θεωρώ, και όλε οι ομάδε, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο διαχωρισμένε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε θέλουμε περισσότερε πληροφορίε, πλήρε πληροφορίε. θέλουμε, είναι άλλοι που λένε ναι, αλλά άμα είναι πάρα πολλέ πληροφορίε, πληροφορίες, μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, ε, Επίτροπε. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα στον τομέα της υγείας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά προνόμια για ζητήματα υγείας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πραγματικά ευχαριστώ πολύ και για τη σαφήνειά σας, αλλά και για τη δέσμευση που έχετε αναλάβει ενώπιον των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω επ' αυτού. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την εναρμονισμένη μεθοδολογία για την ταξινόμηση και την ε, καταγραφή των ε, παραπώνων των καταναλωτών, βλέπω ότι το έχετε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά σας. Είναι διαφορετική όμως η εμπειρία των διαφόρων κρατών μελών σε αυτό το θέμα. Όπω επίση και στο επίπεδο τη προστασία καταναλωτών. Γι' αυτό είμαι υπέρ μια εναρμόνιση ε, των προτύπων προστασία καταναλωτών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Κάτι σε σχέση με τους ασθενείς ε, που είναι επίσης καταναλωτές. Βλέπω επίσης το πρόγραμμά σας μία πρόταση οδηγίας ή κανονισμού για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα. Πρόκειται για κάποιες τεχνικές προσαρμογές ή έχετε σκοπό να προτείνετε Σοβαρότερε αλλαγέ στον τομέα αυτό των ιατροτεχνικών βοηθημάτων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά αυτά τα σημεία που θέσατε, κυρία Γκέπχαρτ. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Κάτι θα ήθελα να τονίσω απλώς. Την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, η οποία λείπει και η οποία δημιουργεί η έλλειψή τη δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνη, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να του δώσουμε κάτι. Και εσεί υποσχεθήκατε ότι θέλετε να το κάνετε αυτό. Δηλαδή κάτι που να μπορεί να εξασφαλίσει στους πολίτες ότι όταν θα έχουν ένα πρόβλημα μπορούν να κάνουν το παραπονό τους και να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης. Αν δηλαδή ψωνίσουν κάτι ε, κάπου αλλού μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας το είπατε κι εσείς ότι θέλετε να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Επίσης θα συμφωνήσω με αυτό που ζήτησε ο κύριος Ροσφόρ. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, διαβουλεύσεις, συζητήσεις. Εντάξει, θέλετε να κάνετε κι άλλη μία, κάντε κι άλλη μία, συμφωνώ. Αλλά μετά αποφασίστε και δώστε μας κάτι συγκεκριμένο για να δουλέψουμε. Πάντα οι προκατοχοί σα το ίδιο έκαναν. Εντάξει, κάποια στιγμή βάλτε και μια τελεία όμως, ε, δηλαδή πάρτε και μια απόφαση για να μπορούμε κι εμείς να δουλέψουμε. Ελπίζουμε αυτό να γίνει μέσα στο 2010. Κύριο Σφάμπ. Όχι. Τότε να δώσω και πάλι το λόγο στον ε, Επίτροπο για να απαντήσει. Αν δεν προλάβετε μπορείτε να μας απαντήσετε γραπτός μέσω των υπηρεσιών σας. I Κοιτάξτε. Ενημερώθηκα για το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Αράιες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και μπορώ να πω ότι θα σας υποστηρίξουμε πλήρως. και για την εξάπλωση αλλά και για τον έλεγχο ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπήρξαν κάποια ζητήματα σε σχέση με το πόση πρόσβαση έχουν οι χρήστες στο διαδικτύο. Θα προσπαθήσουμε να την επεκτείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κατακαιρματισμός, όπως αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας, για τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών στον κόσμο αυτόν του διαδικτύου. Είναι πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει και εμπιστοσύνη Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, ανάπτυξη μηχανισμών κατά της παραποίησης, για παράδειγμα. Δηλαδή, να γνωρίζει κανείς όλες τις πληροφορίες για ένα προϊόν και να γνωρίζουν και οι ασθενείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Να υπάρχει δηλαδή ένα καλό φιλτράρισμα της ποιότητας των πληροφοριών που λαμβάνουν οι πολίτες, οι καταναλωτές. Η ασφάλεια του διαδικτύου για τους ανηλίκους. Και αυτό είναι εξαιρετική σημασία για μας. Πώς μπορούν επίσης οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο καλύτερα. Πιστεύουμε ότι στο βαθμό του δυνατού πρέπει να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιούν οι πολίτες την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, γιατί υπάρχει κάποιο επίπεδο εναρμονισμού. Βέβαια, ξέρω ότι σε μερικέ χώρε, εναρμόνιση, συγγνώμη, ξέρω ότι σε μερικέ ε, περιπτώσει δεν δουλεύει πολύ καλά. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε καλύτερη πρόσβαση των χρηστών, εξασφαλίζοντας ότι γνωρίζουν όπου και αν βρίσκονται τι δικαιώματα έχουν, με την τηλεφόρτωση για παράδειγμα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι επιχειρήσει να χρησιμοποιούν περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε, να γνωρίζει ο επιχειρηματία ότι έχει κάποιε υποχρεώσει. Να ξέρει δηλαδή ο επιχειρηματία, ο καταναλωτή του που θα αγοράσει σε οποιαδήποτε χώρα, τι δικαιώματα έχει και τι υποχρεώσει έχει. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και να δούμε τι στόχους θέλουμε να επιτύχουμε. Πρώτα θα αποφασίσουμε για το στόχο και μετά θα δούμε τι μέθοδο θα ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε το στόχο. Κύριε Γκρέκ. E Είναι γεγονός ότι σήμερα ο καταναλωτής βρίσκεται στην καρδιά όλων των πολιτικών. Και για την ψηφιακή ατζέντα, και για το κλίμα, και για την ενέργεια, και για τις μεταφορές. Ανεξαρτήτως του ζητήματος, ο καταναλωτής είναι το επίκεντρο της προσοχής. Αυτό είναι το δικό μου καθήκον. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε πρωτοβουλία που προτείνεται από τους συναδέλφους μου και από μένα, πρέπει να την αναλύουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη το συμφέρον του καταναλωτή. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό τομέα. Ξέρετε ότι υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια περιορισμού του, του ηλεκτρονικού εμπορίου ορισμένων προϊόντων. Και η ιδέα ήταν να προστατεύσουμε κάποια προϊόντα και κάποιες εταιρείε. Η ιδέα ήταν επίσης κανονισμούς με αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Αλλά εμείς αντισταθήκαμε και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Ο καταναλωτής μέχρι τώρα παρέμενε κάπως αδρανή σε όλα αυτά. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι ο καταναλωτής παραμένει το επίκεντρο της προσοχής στο πλαίσιο της δουλειάς μας. Η συνέπεια του καταναλωτή είναι προτεραιότητα. Βέβαια, η νομοθεσία θα εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικός είμαι εγώ. πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι εμεί συνεργαζόμαστε στην Επιτροπή. Όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία του καταναλωτή. Και δεν νομίζω ότι έχω αντιμετωπίσει προβλήματα συνεργασίας με άλλους συναδέλφου. Τώρα, να τονίσω και πάλι ότι δεν θα ισχύσει αμερικανικού τύπου νομοθεσία. Όχι, σας το λέω κατηγορηματικά, το επαναλαμβάνω και ελπίζω Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Σας το λέω για να ησυχάσετε. Κυρία Γκέπχαρτ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. επιμένουμε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Γκρέκ. Το ανέφερε. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε πολύ, ενδεχομένως ένα μήνα. Αλλά θα επιμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα, να μην ξεφύγουμε από την πορεία μας. Του χρόνου να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι είναι εξαιρετική σημασία. για να μπορεί να, είναι και πάλι, να έχει και πάλι εμπιστοσύνη ο καταναλωτής στην ε, ε, εσωτερική αγορά. όσον αφορά την ε, ανεπαρκή εκπροσώπηση των καταναλωτών. Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό. Εμείς προσέχουμε πάρα πολύ τους καταναλωτές. Χτες Ήμουν στη Ουάσιγκτον. Και μία από, τις, από τους βασικούς λόγους που πήγα εκεί ήταν ο διατλαντικός διάλογος ε, των καταναλωτών στη Ουάσιγκτον. Το κάναμε πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Και τα ακούσματα που έχουμε είναι πάρα πολύ θετικά όσον αφορά την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Ευπρόσδεκτο θα είναι οτιδήποτε μπορείτε να μας δώσετε ως πληροφορία σε σχέση με την οδηγία αυτή. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για ό,τι κάνουμε. Το να συμμετέχει η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίση. Έχω πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Χτε μόλι γυρίσα, σα το είπα συζητήσαμε και αυτό το θέμα. Ελπίζω μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια των προϊόντων. Εγώ τους είπα ότι είναι επωφελές για όλους και μάλιστα πρότεινα να συμμετέχει και ο Καναδάς. Γιατί όχι. Όσο μεγαλύτερο είναι το δίκτυο τόσο περισσότερο προστατεύουμε τους καταναλωτές μας. Γιατί αυξάνουμε και τη δυνατότητα που έχουμε για έλεγχο των προϊόντων. Γιατί με τη συνεργασία αυτή υπάρχει μια ανταλλαγή ελέγχων. Στην Κίνα θα πάω τον Ιούνιο και ένα από τα ζητήματα που θα επιμείνω να συζητηθούν, να συζητηθεί, είναι πώς θα ελέγξουμε την, πηγή, την ε, ποιότητα στην πηγή στην Κίνα. Κοιτάξτε, είναι γνωστό το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Το συζητήσαμε και χθε με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ. Μία κοινή προσέγγιση της Κίνας. Από κοινού, δηλαδή, να ενισχύσουμε την άποψή μας, μιλώντας με την Κίνα. Επίσης, υποστήριξη του προπολογισμού. Στη Μάλτα 10 χρόνια ήμουν Υπουργός Οικονομικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα αιτήματα νέων προγραμμάτων, να, να ε, χρηματοδοτούνται επαρκώς. Διαφορετικά, τα αποτέλεσμα θα είναι μετριότητα. Δεν μιλάω μόνο για τα πιλωτικά προγράμματα. Τα πιλωτικά προγράμματα έχουμε ήδη αρκετά. Το βασικότερο είναι η ανάπτυξη υποδομών. Γιατί όπως γνωρίζετε, ένα μία από τις βασικότερες κριτικές που ακούμε, ακόμη και από εσά από το Κοινοβούλιο, είναι ότι δεν επιβάλλονται οι κανόνες σε πολλού τομεί. Είναι εύκολο για μένα να πω αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αν δεν αυτό το θέμα, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, για να έχουμε αποτελέσματα για του πολίτε μα. Άρα, θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω συνεχώς πάρα πολλέ φορέ θα σα το πω. Δεν θα σα πω ποτέ ότι δεν είναι δική μου ευθύνη. Είναι δική μου ευθύνη και πρέπει να εξασφαλίσω ότι όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο και να οικοδομήσουν το δυναμικό τους έτσι ώστε να μην υπάρχει διάχυση δυνάμεων. Βεβαίως η έλλειψη εποπτείας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, αλλά μιλάμε και για την ε, διατροφική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων γενικότερα, άλλα θέματα υγείας και υγιεινής όπου υπάρχουν ε, ε, επιδημίες και τάσεις επιδημίας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, διότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια για την εναρμόνιση των παραπώνων των καταναλωτών. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε γρηγορότερα στα παράπονα, στις αιτιάσεις των καταναλωτών. Ως προς τα ιατρικά μηχανήματα, τον ιατρικό εξοπλισμό, οι ε, βασικές αλλαγές που θα επέλθουν είναι οι γενετικές δοκιμές, καλύτερη εποπτεία και η ισχύ, θέση σε ισχύ της ποιότητας των ιατρικών αυτών, του ιατρικού αυτού εξοπλισμού. Ευχαριστώ. Uh, John, thank you Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ασχοληθήκατε με ένα τόσο ευρύ φάσμα θεμάτων μεταξύ των οποίων οποίων πολλά που δεν άπτονται της άμεσης αρμοδιότητάς σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Ε, μας δώσατε ένα εντυπωσιακό φάσμα θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας και στον έλεγχό σας και θα ήθελα να σας συγχαρώ, διότι όταν ε, ήρθατε σε αυτή την ακρόαση, η κυρία Γκέμπχαρτ σας ε, υπέβαλε μία συγκεκριμένη ερώτηση, ότι είσαστε ο επικεφαλής των καταναλωτών στην Επιτροπή και αυτό το αποδείξατε μέσα στο ευρύ ε, φάσμα θεμάτων που μας απασχόλησαν από την ε, ηφαιστειογενή λάβα μέχρι θέματα διατροφικής ασφάλειας. Θα, συνεχίσετε, θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας για το υπόλοιπο της θητείας σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναβρεθούμε και θα συνεργαστούμε και χαιρόμαστε που και η ομάδα σας παρευρίσκεται εδώ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Κυρίες και κύριοι, τελικό θέμα που θα μας απασχολήσει. Έχουμε συρρυκνώσει το χρόνο του εισηγητή, γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω κάτι. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση και δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Ο κύριος Ντάλι ασχολείται με το θέμα, αλλά και ο κύριος Κρέτς. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε χρόνο να, το, να την εξετάσουμε πλήρως αυτή την έκθεση και οι σκιώδεις μας έχουν δώσει εντολή να μιλήσουμε στη θέση τους, εν ονόματί τους δηλαδή. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος με την παρουσία των σκιωδών. Θα θέλαμε να σας προτείνουμε λοιπόν στις 2 Ιουνίου Καταρχήν η κυρία Κρός θα έρθει στην Επιτροπή στις 2 Ιουνίου, άρα ίσως να θέλει να σχολιάσει την έκθεση, αλλά μπορούμε να έχουμε και μία ώρα παραπάνω την ε, Τετάρτη το απόγευμα 2 Ιουνίου, έτσι ώστε όλοι να συμμετάσχουν. Διότι η προθεσμία για τις τροπολογίες που δεν είναι ρεαλιστική, γιατί ούτε καν συζητήσουμε είναι η 5η Μαΐου. Εφόσον η Σκιώδης δεν είναι εδώ, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι έκθεση ίδιας ε, πρωτοβουλίας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, προθεσμίες, τις αυστηρές ε, προθεσμίες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι συντονιστές θα ήθελαν να σχολιάσουν Νομίζω θα ήταν καλή ιδέα κάπως να παρεκτείνουμε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα. Οι πολιτικές ομάδες θα ενημερώσουν τους σκιώδεις και θα έχουμε ορισμένα πρωταρχικά σχόλια σήμερα. Αλλά νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ σημαντική και δεν θέλουμε να συρρυκνώσουμε το ε, χρόνο σας. Σας δίνω το λόγο να μας κάνετε μια εισαγωγή. Ευχαριστώ. Ε... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί θα ήταν σκόπιμο να αναβάλουμε την προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το έγγραφο. Καλό σας απόγευμα. Από τότε που ορίστηκα εισηγητής και επειδή μιλάμε για την συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εργάστηκα τους τελευταίους μήνες ε, για το θέμα αυτό, δηλαδή το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και η παρούσα έκθεση είναι απότοκη των μελετών σε σχέση με το εμπόριο online και ε, ήρθα σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώσεις καταναλωτών και γενικότερα εμπλεκόμενους φορείς ε, που θέλησαν να με βοηθήσουν για το εμπόριο online. Κατά τη διαδικασία αυτή είδα ότι ανακύπτουν πολλά προβλήματα τα ε, οποία οδηγούν σε προσκόμματα, έτσι ώστε να μην μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο. Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια κινητήριος δύναμη του διαδικτύου και καταλήτης για να φτάσουμε στους απότερους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Είναι ζωτική σημασίας να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να αρθούν τα, προσκόμενα, τα προσκόμματα με συγχωρείτε, ως προς το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ένας από τους ε, βασικούς ε, παράγοντες για να φτάσουμε στο στόχο αυτό είναι μία διαδραστική πολιτική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί πλήρως το ηλεκτρονικό εμπόριο και να ε, παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες καλής ποιότητας. Έτσι θα μπορέσουμε όχι μόνο να συμπληρώσουμε την εσωτερική αγορά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά να βοηθήσουμε και την εσωτερική αγορά μέσω αυτού. Στην παρούσα κατάσταση χρηματοπιστωτικής κρίσης, το να άρουμε αυτά τα προσκόμματα θα οδηγήσει στην άρση των ανισορροπιών και θα βοηθήσουμε τους ε, πλέον ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα δώσουμε ένα δυναμικό χαρακτήρα στην οικονομία μας. Θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο για όλους τους πολίτες και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε αποτελεσματικές ε, πολιτικές έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την δυναμική πορεία της αγοράς. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς που αποτελούν πρόσκομα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην πλήρη ανάπτυξή του. Όπως σας είπα, στις 17 Μαρτίου χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αγορά η οποία να είναι δυνατή και εύρωστη έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί προς το εξωτερικό. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικές προς τα έξω. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί ανά τον κόσμο, για να ακολουθήσουμε το μονοπάτι ενός πραγματικού ε, ηλεκτρονικού εμπορίου και ανταγωνιστικότητας παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα είναι γεμάτη από προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε παγκόσμια κλίμακα. Το διαδίκτυο και οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες οδήγησαν σε μια επανάσταση χωρίς προηγούμενο. Δεν μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας αν δεν αναπροσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα. Όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία. Θεωρώ ότι έξι είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Εκεί επικεντρώνω την προσοχή μου. Θα πρέπει να υπάρχει ε, ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι καταναλωτές χρειάζονται μία ποιοτική πρόσβαση στο δίκτυο, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών και να αυξηθεί η ποιότητα και η ταχύτητα ενδοκινοτικά τουλάχιστον για αυτούς που δεν έχουν καλή διαδικτυακή πρόσβαση. Επίσης, πολλοί πολίτες δημιουργούν προσκόμματα διασυνοριακά και δεν υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες για ορισμένες περιφέρειες, είτε διότι δεν πολλούν σε καταναλωτές ορισμένων χωρών. Άρα χρειάζεται μεταξύ άλλων μέτρων να ενισχύσουμε την εφαρμογή του άρθρου 20 σημείο 2 που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την υπηκότητα ή την ηθαγένεια. Θα πρέπει να υπερβούμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Αυτό θα είναι ένα βασικό βήμα, όχι ε, κατά τη σύναψη συμβάσεων, αλλά και για να επιλύσουμε προβλήματα τα οποία θα μπορέσουν να ανακύψουν μεταξύ αγοραστή και πολιτή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όταν αγοράζουν online. Μερικοί καταναλωτές δεν αγοράζουν online διότι δεν πιστεύουν στην ασφάλεια αυτής της αγοράς. Για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να προωθήσουμε συγκεκριμένες δράσεις. Να εφαρμόσουμε ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό σήμα όσον αφορά, την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να είναι σίγουροι ως προς την ε, καταβολή της ε, πληρωμής online, δηλαδή για την ασφάλεια της πληρωμής. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για να ζητήσουμε από τους επιχειρηματίε να θέτουν σε εμπορία τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. Πολλοί δεν το κάνουν, διότι υπάρχουν ε, πολλά μειονεκτήματα ως προς τη φορολόγηση ως προς την διαχείριση αποβλήτων και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μεγάλες λοιπόν διαφορές γι' αυτό. Ε, πρόκειται για ένα δαπανηρό και πολύπλοκο εγχείρημα. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπουν σε αυτήν η μειοψηφία να πολύ online. Και αυτό αφορά και τον μηχανισμό καταβολής ΦΠΑ την εναρμόνιση των δαπανών όσον αφορά τα ταχυδρομικά τέλη ή τα τραπεζικά τέλη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να καταβάλουν ένα αντίτιμο σε διάφορες χώρες για την ίδια υπηρεσία οι καταναλωτές και να μην, υπάρχουν, ε, ε, ε, να μην υπάρχει ρήξη μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, ρήξη συμφερόντων θα πρέπει να υπάρξει ασφάλεια ως προς τους ανηλίκους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας των ανηλίκων και να προωθηθούν εκστρατείες πληροφόρησης προς τους γονείς, τους καθηγητές και τους κηδεμόνες, έτσι ώστε να γνωρίζουν την ευθύνη τους στην εκπαίδευση των ανηλίκων ως προς την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ΙΜΚΟ, διότι ήταν διαθέσιμη και άκρος επαγγελματική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, διότι ήταν διαθέσιμοι με υποδείξεις κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων των τελευταίων μηνών. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των μελών αυτής της Επιτροπής, καθώς και τις υποδείξεις της Επιτροπής, που είδα ότι είναι παρούσα και άλλων ενδιαφερομένων και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις πριν από την τελική έκβαση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ράιος για, το, για την εισαγωγή αυτή. Δύο επιτροπές θα χνομοδοτήσουν, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Οπότε, ελπίζω ότι το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα θα βοηθήσει και αυτές τι επιτροπές. Κύριε Σιβίτσου, εσείς είστε εισηγητή στι άλλες ε, επιτροπές. Υποθέτω πως ναι. Καλώς ήρθατε. Είστε ούτω ή άλλω ένα πληρωματικό μέλο τη επιτροπή μας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιοριστώ γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να πατήσετε το μικρόφωνο, γιατί διαφορετικά δεν εμφανίζεστε ε, στο, στο web streaming. Μάλλον είναι το άλλο μικρόφωνο αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Ναι, συνήθως κάθομαι από την άλλη μεριά, γιατί εκεί είναι η πολιτική μου ομάδα. Έλεγα ότι είναι κάποιο είδου διάκριση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα όμω κοιτάξτε, εμφανίζεστε σε, σε full screen, ολόκληρη την οθόνη. Πιάνετε. Πώ σα φαίνεται αυτό. Μουβίμε Κοιτάξτε, είναι πραγματικά επαναστατικό αυτό το ζήτημα. Είναι, μερικά, είναι από τα ζητήματα που λίγες φορές έχουν, ε, τα έχουμε δει στην ιστορία. Είναι πραγματικά μία επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αγοράζονται τα ε, προϊόντα. Είναι συναρπαστικό αυτό το θέμα και όταν είναι συναρπαστικό το θέμα, συνήθω δεν έχουμε πάρα πολλέ γνώσει γι' αυτό. Είμαστε πολύ ενθουσιώδει για να μάθουμε περισσότερο, περισσότερα. Συχνά λοιπόν δεν έχουμε αρκετέ γνώσει για αυτό το θέμα. Και αυτό ισχύει και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγώ διάβασα την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι υπάρχουν μερικές παγίδες που δεν τις αποφύγαμε σε σχέση με την απλοποίηση. 100 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το δυναμικό αυτής της αγοράς. Αλλά μην πέσετε σε αυτή την παγίδα του υπερενθουσιασμού. Αν αγοράσει κανείς ένα ψυγείο στο διαδίκτυο, σημαίνει ότι δεν θα το αγοράσει κανεί σε ένα παραδοσιακό κατάστημα. Κερδίζει στο διαδίκτυο, χάνεις αλλού, σε ένα πραγματικό κατάστημα, στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν λίγο προσεκτικοί γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο επί καθημερινής βάσεως. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν με τις ε, υπερβολικά ενθουσιώδεις προσεγγίσεις μας. Ορισμένα ακόμη σχόλια που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και δεν το κάναμε ή το κάναμε αλλά εν μέρη. Μιλάμε για πιο ανοιχτό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, γιατί στο σημείο που θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτό είναι τελικά περιορισμένο. Γιατί, γιατί κάποιοι πελάτες, κάποιοι καταναλωτές την χάνουν διακριτικής μεταχείρισης. Έχουμε και οδηγία που λέει ότι απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση. Αλλά εγώ είμαι κάτοχος πολωνικής πιστοτικής ε, ε, ε κάρτας, αλλά δεν μπορώ να αγοράσω στο διαδίκτυο κανένα προϊόν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν αναγνωρίζεται η κάρτα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους καταστηγματάρχες. Πάρα πολύ καλό είναι λοιπόν να έχουμε ωραίες ιδέες, αλλά να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι και να τα βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά πρώτα η διακριτική μεταχείριση και μετά συζητήσουμε τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγγύησεις, ε, δυνατότητες ε, ε, αποκατάστασης ζημιών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και δικαίω ο εισηγητή αναφέρει ότι οι καταναλωτέ ακόμη δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδου αγοραπολισίε, γιατί δεν μπορούν να πάρουν στα χέρια τους ένα, όντο, ένα προϊόν, το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λοιπόν αγοραπολισίας. Καλό είναι αυτό να το αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν και σε ένα κανονικό μαχαζί. Αν αγοράσει κανείς ένα πλυντήριο πιάτων ή ένα ψυγείο στο διαδίκτυο, πρέπει να μπορεί να το επιστρέψει αν είναι λατωματικό να το αντικαταστήσει αν δεν λειτουργεί καλά. Κάποιοι φοβούνται, δεν το τολμούν. Γιατί νομίζουν ότι άμα αν αγοράσω ένα ψυγείο στο διαδίκτυο, τι θα κάνω μετά αν δεν δουλεύει καλά. Οπότε καλύτερα πάω σε ένα παραδοσιακό κατάστημα. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αξιοπιστίας ε, ε, ε, πολιτών, εμπόρων, που είναι κάτι το οποίο στην περίπτωση των παραδοσιακών καταστημάτων έχει χτιστεί με τα χρόνια. Το ίδιο πρέπει να πούμε και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλοι όσοι πολλούν διαδικτυακώς πρέπει να οικοδομήσουν αυτήν την αφοσίωση στους καταναλωτές, στους πελάτες τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν τα κίνητρα οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ε, ε εμπόριο. Κοιτάξτε, αν μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα πολύ σαφές ε, σύστημα επίλυσης διαφορών, τότε οι αγοραπολισίες μέσω του διαδικτύου θα επιτύχουν. Πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων και των διαφορών κάτι σαν δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, όπως... Ε, ποιος έχει έναν συγκεκριμένο τομέα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό ε, επί του θέματος αυτού, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Δίκιο έχεις που μας τα υπενθυμίζεις όλα αυτά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τμήμα της ε, γενικής αγοράς. Το να συμπληρώσουμε τα κενά του ηλεκτρονικού εμπορίου σημαίνει ότι συμπληρώνουμε τα κενά που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά γενικώ. Δεν είναι ανεξάρτητα τα δύο πράγματα. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά μήπως... Ε, ποιος είναι ο κύριος David Mayer. Ένα μικρό σχόλιο να κάνω κι εγώ, σύντομο σχόλιο. Πρώτα η κυρία Στήλερ. Uh, right. Well, that's fine then. Okay. Well, um, well, I, I think you have a choice actually. Um, I was going to just invite the Commission to set the scene. Θα καλούσα την Κομισιόν καταρχήν να απαντήσει, εκτός αν θέλετε να μιλήσετε τώρα ή αν θέλετε να κόψουμε την κουβέντα εδώ και να τη συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση και η κυρία Γκέπχαρ θέλει να μιλήσει. Μήπως λοιπόν να μιλήσετε εσείς πρώτα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκέπχαρντ να μιλήσει πρώτη. Όχι, η κυρία Στήλερ θα μιλήσει πρώτη. Σύντομα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς έχει εκτοξευθεί το επίπεδο των, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλο και περισσότεροι ψωνίζουν ε, χριστουγεννιάτικα δώρα online. Γι' αυτό και η Amazon έγινε τεράστια επιτυχία. Και φέτος Έκλεισαν και κάποια μαγαζιά λόγω των, ε, καταστήματα λόγω των ε, εμπορικών συναλλαγών στο ίντερνετ. Τώρα μπορεί κανεί να έχει και κάθε τα περισσότερα μάλλον καταστήματα έχουν και στο σελίδε και μπορεί κανεί να αγοράσει τα ηλεκτρικά του, ε, τι ηλεκτρικέ του συσκευέ, ε, τα πάντα στο ίντερνετ. Βεβαίω εδώ πρέπει να υπάρχει σημαντική πτυχή τη ε, προστασία των καταναλωτών και βεβαίω εδώ έχουμε να κάνουμε και με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτοί που αγοράζουν στο ίντερνετ δεν είναι φτωχό συγγενείς. Οπότε έχουμε πολλέ ευκαιρίε εδώ και πολλέ δυνατότητε. Ευχαριστώ για τον, τον εισηγητή λοιπόν για τη δουλειά που έκανε και τι απόψει που παράθεσε στην ε, έκθεση. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Γιατί ο συνάδελφος μου έδωσε τη σημειώση στα γαλλικά γι αυτό, και γι' αυτό θα μιλήσω στα γαλλικά. Ε, είναι δύο γεμάτες σελίδες Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, αναφέρω σημεία, ορισμένα σημεία, να, αναφέρω ορισμένα σημεία για τον κύριο Αρίας. Σας ευχαριστώ για αυτό το πολύ χρήσιμο κείμενο το οποίο αναφέρεται στα εγγενή προβλήματα αυτής της πλευράς της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία είναι ύψη τη σημασίας και πρέπει να υπογραμμιστούν και είναι ιδιαίτερα θετικά. Υπάρχουν και ορισμένα σημεία που ίσως ανακύπτουν ορισμένα προβλήματα και χρειάζεται κάποια συζήτηση. Δηλαδή, ως προς το παράδειγμα που επιλέξατε, γιατί λέτε ότι τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών ενδιαφέρονται για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς. Συμφωνώ μαζί του ότι ε, δυστυχώς ότι συμβαίνει το αντίθετο. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να υπηρετεί τον καταναλωτή. Στο σημείο 4 ε, γίνεται μνήα στα λεγόμενα της Επιτρόπου Ρέντινγκ ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να κινηθούμε. Στο σημείο 14 γίνεται λόγος για το κατά πόσο χρειάζεται να συντάσσονται τόσοι κανονισμοί και στο σημείο 19 κατά πόσο είναι αναγκαίο να δημιουργούμε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την προστασία του καταναλωτή ή δεν υπάρχουν άλλα μέσα για να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Ίσως θα πρέπει να δούμε καλύτερα το θέμα των πληρωμών online. Ο κύριος Σίβετς είπε ακριβώς αυτό. Είναι επίσης ύψης της σημασίας. Στο σημείο 25 προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος επιδοτήσεων και ο συνάδελφος και εγώ πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν ε, ιδιαίτερα αποδοτικό. Ίσως θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο με σαφείς κανόνες για το ΦΠΑ, πνευματική ιδιοκτησία, σύστημα πληρωμών και ταχυδρομικές υπηρεσίες σε δίκαιες τιμές, παρά να γίνονται επιδοτήσεις. Αυτή, αυτή ήταν η ουσία ε, αυτών που μου ανέφερε ο συνάδελφος. Ήθελε και άλλα σημεία να αναφέρει, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι η βάση αυτών που προτείνατε, κύριε Αρίας, είναι μια πολύ καλή βάση, ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης και θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Good. Uh, thank you very much Ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο. Οπότε ας δώσω το λόγο στον κύριο Μέιρ να σχολιάσει για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες της Κομισιόν, ειδικά για την ε, αλυσίδα διανομής. Τροφοδοσία, συγγνώμη. Η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα ε, ενέκρινε μία σχετική πρωτοβουλία Αναφέρεται και στην ε, έκθεση βεβαίω του κυρίου Αρίας, αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε. Οι συνάδελφοι από την ΕΚΟΝ λένε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι σημαντικά στην, ε, για τους ε, καταναλωτές και πρέπει να συζητούνται πιο γενικόλογα. Μήπως μπορείτε λοιπόν εσείς να μας κάνετε ένα σχόλιο. Um, how this is going to move forward. Ευχαριστώ. Νομίζω θα είμαι σύντομος. Γιατί ούτως σύντομο. έδωσε εκτενή απάντηση στον κύριο Αρία. Απλώ θα επιβεβαιώσω ότι η αλλω ο επιτροπο σανταλη εδωσε εκτενη απαντηση στον κυριο αριας απλως θα επιβεβαιωσω οτι η πτυχη των καταναλωτών στο θέμα που θίξατε είναι πολύ σημαντική. Και τα μελετούμε τα θέματα αυτά εντελεχώς. Και βεβαίω η συμβολή του Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντική στη δουλειά που κάνει η Κομισιόν φέτο. Uh, Ειδικά για τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ευχαριστώ. Αξιοθαύμαστη η συντομία σας. Θα σας έχω υπόψη μου και για το μέλλον. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο πιο λεπτομερές ε, χρονοδιάγραμμα μετά τις 2 του Ιούνιου για, την, ε, για να ψηφίσουμε την έκθεσή σας μάλλον ε, τον ε, Σεπτέμβρη, γιατί έχουμε και δύο συνόδους ολομέλειας τότε. Οπότε να δώσουμε τώρα το, το λόγο στον κύριο Αριάς για να σχολιάσει. Ο κύριος Σίβιτς, είστε ο συγητής γνωμοδότησης για άλλη επιτροπή. Όχι, δεν είστε τίποτα. Πολύ ωραία. Εντάξει, από μόνο σας ήρθατε. Πολύ ωραία. Οπότε μή, μήπως θέλετε να κάνετε μια, άλλη, μια γνωμοδότηση για μια άλλη επιτροπή. Δεν πήρατε καμιά ιδέα σήμερα. Ο κύριος Αρίας έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ το σχόλιο σε σχέση με ε, τις τροπολογίες προθεσμία 2 Ιουνίου. Αυτό είπατε? Όχι. Θα ορίσουμε νέα προθεσμία. Θα το ξανασυζητήσουμε την έκθεσή σας στις 2 Ιουνίου και θα έχουμε και την παρέμβαση της Επιτρόπου Κρούς και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί όλα αυτά διασυνδέονται. Και θα το δούμε και με τις Επιτροπές ε, Γνωμοδότησης, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα προθεσμία αργότερα τον Ιούνιο. Άρα θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο και σε μία από τις δύο συνόδους του Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει η Ολομέλεια. Άρα έχετε αρκετό χρόνο. Μετά θα συνεργαστούμε με τις επιτροπές που γνωμοδοτούν επίσης. Ωραία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν σήμερα για την έκθεση αυτή και να πω ότι καταγράφω τα όσα είπαν και βεβαίως θα συζητηθούν και εφόσον παρεκτείναμε την προθεσμία νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο, να, με απασχολήσουν περισσότερο τα σχόλιά σας και οι υποδείξεις σας. Και επειδή πέρασε και η ώρα, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσω εδώ. Well, thank you very much Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι και εσείς και οι σκιώδεις θα χρησιμοποιήσετε το χρόνο εύλογα. Ωραία. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 10 Μαΐου θα συνεδριάσουμε από τις 3 μέχρι τις 6.30 ε, έτσι ώστε να δούμε την τότε ημερήσια διάταξη και στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε πάλι συνεδρίαση της Επιτροπής με δύο συνεδρίες. Αναμένουμε και την κυρία Κρούς ε, ε, στην Επιτροπή. Θα τα πούμε τότε. Σας ευχαριστώ και να σας χαιρετήσω. Χαίρετε λοιπόν.